Ladies and gentlemen. Good Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στο δεύτερο τμήμα της ε, εκδήλωσης που προβλέπει το συνδυασμό της εργασίας με την ζωή εκτός εργασίας, ε, βιώσιμη απασχόληση κατά τη διάρκεια της ζωής. Ονομάζομαι Μάρια Χάκινγκ, θα είμαι η πρόεδρος σήμερα και έχω και ε, πολύ σημαντικούς καλεσμένους, τους οποίους θα παρουσιάσω σε λίγο. Ε, ξεκινάμε μια καθυστέρηση, αλλά μετά θα είμαστε πολύ πιο αυστηροί στην τήρηση του χρόνου. Θα είμαι λακωνική, δίνοντας το καλό παράδειγμα. Τι εξετάζουμε σήμερα. Την προσέγγιση του κύκλου της ζωής, που είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Κάποτε πίστευα ότι είναι πιο σημαντικό αυτό για τις γυναίκες παρά για τους άντρες ιδιαίτερα γιατί φροντίζουν οι γυναίκες ε, άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτά τα πράγματα όμως αλλάζουν, οπότε η προσέγγιση που θα υιοθετήσουμε στον τομέα αυτό, όποια και αν είναι, θα πρέπει να είναι ουδέτερη από άποψη φύλου. Τι έχουμε ενώπιον μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν, γονική άδεια. Εκεί περιμένουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, ε, για την ισορροπία εργασία και προσωπική ζωή. Ο πρόεδρο Γιούνκερ μα μίλησε για τον πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και ευελπιστώ ότι στην ανακοίνωση αυτή για την ισορροπία ε, εργασία ε, και προσωπική ζωή θα δούμε κάτι και για όσου επιφορτίζονται τη φροντίδα των άλλων μελών τη οικογένεια. Μάλιστα, πήγα σε μια διάσκεψη στη Σλοβενία την προηγούμενη εβδομάδα και εξετάσαμε αυτό το θέμα, αλλά από την προοπτική των συντάξεων περισσότερο από την επάρκεια και κυρίως τη βιωσιμότητα των, των συντάξεων από αυτή τη σκοπιά. Επίσης, έχουμε και το θέμα της ε, εργασίας ε, και της υγείας, υγείας στον χώρο εργασίας. Και εκεί θέλουμε συνέργειες. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις αναντιστοιχίες των δεξιοτήτων, ε, νέα κατάρτιση των εργαζομένων. Μόλις θετήσαμε την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ κάτι που προϋποθέτει τήρηση κάποιων υποχρεώσεων. Επίσης, ε, η πάταξη των διακρίσεων και το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας. Ε, ε, Αξιοπρεπή αμοιβή για, για την εργασία, το κατώτατο εισόδημα πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το μέτρο για να προλάβουμε την ε, φτώχεια. Επίσης, προκλήσεις της ψηφιακής κοινωνίας. Σήμερα το πρωί έκανα μια μιλή σε μια διάσκεψη για γυναίκες επιχειρηματίες ε, που απασχολούνται κυρίως στον τομέα των, πληροφοριών, των, τεχνολογιών κοινωνία, της πληροφορικής και της τεχνολογίας. Θέλουμε ελαστικότητα και αυτό περιέχει η ψηφιακή κοινωνία, αλλά ε, συνεπιφέρει αβεβαιότητα και επισφάλεια. Και επειδή ε, είμαστε άνθρωποι, ανθρώπινα πλάσματα με μια λογική καρδιά, θα πρέπει να δούμε τις συνέπειες ε, αυτής της ε, ψηφιακής κοινωνίας. Οπότε και το θέμα του φόρτου εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε υπό τη σκοπιά αυτής της ανάγκης για αξιοπρεπή απασχόληση. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον συνάδελφο Όλε Κρίστενσεν, που είναι μέλος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από τη Δανία και από τα πιο ενεργά μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης. Α, συγγνώμη. Ε, τρέχω πιο μπροστά και από μένα την ίδια, όπως λέμε και στην Ιλλανδία. Ξέχασα την παρακαθήμενη εξεβονίμων, την Greet Vermeilen, που είναι manager προγράμματος για τις εργασιακές συνθήκες και τις βιομηχανικές σχέσεις από τη Eurofound και προηγείται στην ομιλία. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα στην παρουσίασή μου να σας δείξω κάποιες διαφάνειες και θα εξετάσω κάποια θέματα που θα τα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα και που αφορούν... Ε, το πρωί μιλήσαμε για την ποιότητα της απασχόλησης, τώρα θα δούμε τη διάδραση εργασίας και εργαζόμενου και πώς αυτή η διάδραση, η αλληλεπίδραση εντάσσεται στη διάρκεια της ζωής. Θα δούμε την βιωσιμότητα της ε, εργασίας, ένα κόνσεπτ της Eurofound, ε, την, ε, τον αντίκτυπο της υγείας στην εργασία, τον συνδυασμό της εργασίας και της προσωπικής ζωής και κάποιες παρατηρήσεις και για την ισότητα των φύλων. Η δική μας προσέγγιση για μια βιώσιμη εργασία καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής έχουμε δύο βασικές ε, έννοιε. Καταρχήν πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή περισσότερων ανθρώπων στην ε, αγορά εργασία. Θέλουμε μια περιεκτική, χωρί αποκλεισμού αγορά εργασία ε, να συμπεριλάβει και του σημερινά άνεργους ή για κάποιου που έχουν προβλήματα υγεία, για παράδειγμα. Επίση, θα πρέπει να φροντίσουμε ο κόσμο να είναι ικανό και πρόθυμο να εργαστεί μέχρι την ηλικία τη συνταξιοδότηση, ακόμη και μετά από τη σύνταξη. Επίσης, ε, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις τους προσωπικούς πόρους ό,τι αφορά τις δεξιότητες, την υγεία, ώστε να μπορούν οι συνάνθρωποι μας να εργάζονται μέχρι βαθιά γεράματα. Και επίσης να επικεντρωθούμε στις συνθήκες που επιτρέπουν τον καλύτερο συνδυασμό εργασίας και προσωπικής ζωής. Ε, είτε θα μπορούσαμε να έχουμε μια προληπτική προσέγγιση, η προορατική, και να δούμε πώς ε, μερικές ε, ιδιαίτερες καταστάσεις ή προβλήματα μπορούν να ληφθούν υπόψη ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ε, την εργασία τους οι εργαζόμενοι. Επόμενο θέμα. Δύο στοιχεία, εργασία και ποιότητα εργασίας. Σήμερα το πρωί η Ανιές μας έκανε μια παρουσίαση και μετά είχαμε εκτενή συζήτηση στο πάνελ ε, εκεί διαπιστώσαμε ότι οι καλέ εργασιακέ συνθήκε και η ποιότητα τη εργασία έχουν θεμελιώδη σημασία για να μπορούν οι εργαζόμενοι να συνεχίσουν να δουλεύουν καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Και αυτό γίνεται είτε με πολιτικέ, με νομοθεσία, με συλλογικέ ε, συμφωνίε και πρακτικέ στου χώρου εργασία. Αυτό το συζητήσαμε εκτενώς στο πρώτο τμήμα του σεμιναρίου. Κάποια στοιχεία θα τα δούμε και τώρα, αλλά Τώρα θα ασχοληθούμε περισσότερο με τον εργαζόμενο ώστε να μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Δηλαδή θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαίτερες ε, ε, συνθήκες του εργαζομένου και δεχόμενα ζητήματα που θα ανακύψουν. Επίσης, εξετάζουμε εργαζόμενους κάθε ηλικίας, ε, κάποια θέματα υγείας και γι' αυτό θα πρέπει η εργασία να, να προσαρμόζεται στα θέματα της υγείας. Θα πρέπει να διευκολύνεται επίση από πολιτικές, από κάποιες επιδοτήσει ενδεχομένω ε, και θέματα που θα τα διαπραγματευτούν οι κοινωνικοί εταίροι και ε, θέματα υγείας μπορεί να αφορούν την εργασία αλλά να είναι και άσχετα, για παράδειγμα μια αναπηρία. Θα πρέπει να φροντίζουμε λοιπόν ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να επιστρέφουν στην εργασία τους όποτε, όποτε γίνεται. Επίσης, ευθύνες παροχής φροντίδας, ε, είτε για τα παιδιά είτε για τα εγγόνια ή άλλους, ε, άλλα εξαρτημένα μέλη της οικογένειας, ανάπηροι συγγενείς, ε, ο σύντροφος ενδεχομένω ή ηλικιωμένοι γονείς και αυτό μπορούμε να το επιλύσουμε με διάφορου τρόπου. Θα επικεντρωθούμε κυρίω σε πρακτικέ και ρυθμίσει στο χώρο εργασία, ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι να συνδυάζουν την εργασία με την προσωπική του ζωή. Αυτό όμω που είναι πολύ σημαντικό και θα συζητηθεί επίση αργότερα, είναι κάποιε ρυθμίσει για την άδεια, άδεια γονική, άδεια αυτού που παρέχει φροντίδα. Ήδη άλλες διευκολύνσεις όπως βρεφονιπιακή σταθμή, ε, φροντίδα μετά το σχολείο ή ρυθμίσεις για να προσφέρονται πλέον βοήθεια σε αυτούς που παρέχουν, μεριμνούν για κάποιους ε, συγγενείς τους. Επίσης, οι ανάγκες ε, δεν είναι ίδιες και άρα οι δεν μπορεί να είναι ίδιες. Μείωση του ωραρίου εργασία θα μπορούσε να είναι μια καλή ρύθμιση για να ληφθούν υπόψη επιμέρου προβλήματα πέραν των αδειών. Επίση, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Γιατί άλλη φροντίδα για τα ανήλικα παιδιά και άλλη φροντίδα που χρειάζονται οι ηλικιωμένοι γονεί, για παράδειγμα. Για του οποίου ε, θα πρέπει να βγείτε να κάνετε ψώνια ή να του πάτε σε ένα γιατρό. Διαφορετικέ οι ανάγκε και άρα διαφορετικέ λύσει θα επιλέγονται ανάλογα σε τη φάση ζωή βρίσκεται ο καθένα. Επίσης, συνδυασμός εργασίας και προσωπικής ζωής. Η απασχολησιμότητα όταν χάνει κανείς ε, την ε, δουλειά του, όταν θέλει να αλλάξει δουλειά, πώς μπορεί να αναβαθμίσει τις δεξιότητές του. Επίσης, τι κίνητρα θα πρέπει να δοθούν. Επόμενη διαφάνεια, την, έκθεση για, την έκτη έκθεση για τις εργασιακές συνθήκες. Τι γίνεται με το γεράσκοντα πληθυσμό, το, το εργατικό δυναμικό. Φυσικά θα πρέπει να φροντίσουμε για τις σωστές εργασιακές συνθήκες όλων των εργαζομένων και για να προσαρμοστούμε σε ένα γεράσκον εργατικό δυναμικό θα πρέπει να δούμε τις εργασιακές συνθήκες ε, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, όχι μόνο ε, όσο μεγαλώνουν. Επίσης θα πρέπει να δούμε ε, τους νέους εργαζόμενους που εκτίθεται περισσότερο σε κάποιους ε, σωματικούς κινδύνους. Άλλοι κίνδυνοι ε, απειλούν καθ' τη διάρκεια της ζωής, περισσότερο προς τις μεταγενέστερες φάσεις, βραδινές βάρδιες, βάρδιες γενικώ με ένταση εργασίας. Οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν λιγότερη πρόσβαση στη κατάρτιση, λιγότερες επαγγελματικές προοπτικές, σταδιοδρομία και εκμάθηση. Οπότε όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αν θέλουμε οι εργαζόμενοι να παραμένουν στην εργασία τους περισσότερα χρόνια. Στην έκθεσή μας βλέπουμε ότι 73% των εργαζομένων ε, ισχυρίζονται ότι μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ή κάποια παρόμοια μέχρι τα 60. Και αυτοί που είναι πάνω από 55 θα τους ρωτήσουμε μετά από 5 χρόνια. Δηλαδή, 27% των εργαζομένων ισχυρίζονται ότι δεν είναι σε θέση να διεκπαιρεώσουν τη δουλειά τους μέχρι τα 60. Παρά μόνο μέχρι τα 60 μάλλον. Και ίσως και νωρίτερα. Βέβαια, περισσότεροι άνδρες ε, κάνουν αυτόν τον ισχυρισμό ότι μέχρι τα 60 είναι ικανοί να δουλεύουν και αν δούμε ε, το χάσμα μεταξύ των φύλων δεν είναι πολύ μεγάλο στις διάφορες χώρες. Αν βλέπουμε τους εργαζόμενους που των 25, βλέπουμε ότι είναι μεγαλύτερο το χάσμα των φύλων. Φτάνει και μέχρι τις 20 ποσοστιαίες μονάδες σε μερικέ χώρες. Τώρα, ποιο είναι το θετικό μήνυμα. 80% των εργαζομένων 18% των εργαζομένων λένε ότι θα ήθελαν να δουλεύουν μέχρι τέλος σχεδόν, όσο περισσότερο γίνεται, αν είναι δική τους επιλογή. Και επίσης, ε, ποιοι είναι οι λόγοι που θέλουν να δουλεύουν όσο περισσότερο γίνεται. Όχι μόνο οικονομική, αλλά και κοινωνικού πλαισίου. Θέλουν να, να προσφέρουν στην κοινωνία, να έχουν δουλειά σημαντική που θα τους δίνει κάποιο νόημα. Επίσης, για τις, τους παράγοντες ε, ποιότητας, τους δείκτες ποιότητας πέραν των αμοιβών, βλέπετε τις μπλε στήλες, καλά, καλά είναι τα αποτελέσματα εδώ βλέπετε ότι η βιώσιμη απασχόληση συνδέεται με όλους τους δείκτες ποιότητας της εργασίας και έχει πολύ θετική απήχηση. Επίσης, όταν είναι κακοί οι δείκτες, είναι κακή η επίδραση Επίσης, έκθεση σε σωματικούς κινδύνους, ε, ένταση εργασίας, βάρδιες, ε, νυχτερινή βάρδια, φόβος ε, της απώλειας της θέσης εργασίας, η άδικη μεταχείριση, η παρενόχληση ή το bullying, ο εκφοβισμός, όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα εργασίας και κάνουν πολύ πιθανή την άρνηση το ατόμου να δουλεύει μέχρι τα 60 και επίσης η αναγνώριση που λαμβάνει κανεί στην εργασία του και ε, να μπορεί να φροντίσετε προσωπικά του θέματα ή να βοηθήσει κάποια μέλη της ε, οικογένειάς του. Αυτό δίνει θετικές απαντήσεις όταν υπάρχει θετικό κλίμα. Επίσης, έχουμε εδώ τη χαρτογράφηση των χωρών με τα αποτελέσματα ένα χώρα. Όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα μιας χώρας, τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό των εργαζομένων που ισχυρίζεται ότι είναι βιώσιμη η απασχόλησή τους. 73% των εργαζομένων είπαν θα μπορούσαν να δουλεύουν μέχρι τα 60%. Πάνω από 80% των εργαζομένων στη Γερμανία, Πορτογαλία, Δανία, Σουηδία, Ιταλία και Ιρλανδία ε, και λιγότερο από το 60% των εργαζομένων στην Τουρκία, Γαλλία, Σλοβενία, Ε, ισχυρίζονται ότι θα μπορούσαν να δουλεύουν μέχρι τα 60. Τώρα, ποιότητα ζωής και υγεία. Ποιότητα εργασίας, συγγνώμη, και υγεία. Η σχέση μεταξύ της ποιότητας ε, ζωής και της υγείας είναι πολύ περίπλοκη και αμφίδρομη. Δηλαδή μπορεί να επηρεάζει και τις εργασιακές συνθήκες στην υγεία, αλλά μπορεί να επηρεάζει και την κατάσταση υγείας των εργαζομένων στη δουλειά που μπορούν να κάνουν. Και συνήθως ε, είναι μεταγενέστερα τα αποτελέσματα στην υγεία και μερικοί μπορεί να αποσύρονται νωρίτερα από την αγορά εργασία γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και ίσω και χάσουμε μερικούς εργαζόμενου. Αυτό επηρεάζει την ικανότητά τους να συνεχίσουν να δουλεύουν, αλλά ε, υπονομεύει και την ανάγκη μιας αγοράς εργασίας χωρίς ε, αποκλεισμούς. 26% είναι οι εργαζόμενοι που θεωρούν ότι επηρεάζονται αρνητικά, 28% των ανδρών, 24% των γυναικών, 6% των εργαζομένων έχει κάποιο κίνδυνο να αντιμετωπίσει ψυχικά προβλήματα, ψυχικές ευημερίας, ε, μειοσκελετικά προβλήματα, ποροκεφάλους, κόπωση, πόνο της πλάτης. Επίσης, ε, συμπερίληψη εργαζομένων με χρόνιες νόσους. Περίπου 20% του εργατικού δυναμικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι έχουμε μια χρόνια νόσο που διαρκεί πάνω από 6 μήνες, κάτι που ισχύει περισσότερο για τους ηλικιωμένους, πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, 12% ε, κάτω το 45% και 60% 45% με 59% και ένα στους τέσσερις άνω των 50% ε, ισχυρίζονται ότι έχουν χρόνιες νόσους. Και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη ε, για, αν θέλουμε να παραμένουν πιο πολύ χρόνο στην εργασία οι εργαζόμενοι. Επίσης, είναι σημαντικό και το ρόλο εργασίας ε, να ανταποκρίνεται στο, στην κατάσταση της υγείας. Ένα στους τέσσερις λένε ότι θα χρειαστούν περισσότερες τέτοιες προσαρμογές και ρυθμίσεις στο μέλλον. Τώρα, για να δούμε τους δείκτες. Στα δεξιά έχουμε τους θετικούς και στα αριστερά τους αρνητικούς. Το πορτοκαλί είναι αρνητικό, το γαλάζιο, το μπλε είναι θετικό. Πέραν των δεξιοτήτων και της ε, διακριτικής ευχέρειας έχουμε και το κοινωνικό περιβάλλον στην εργασία. Ε, εκεί περισσότερο έχουμε πανοκεφάλους και προβλήματα ύπνου. Ε, όταν έχουμε περιβάλλον φυσικό περισσότερα έχουμε σωματικά προβλήματα όπως πόνο στην πλάτη, μια σκελετικά και κόπωση Σε ό,τι αφορά την, την ένταση εργασίας, εκεί τα προβλήματα αφορούν περισσότερο δυσκολίες στον ύπνο και μερικά από τα άλλα. Και τώρα κακές προοπτικές, φόβος να χάσει κανείς τη δουλειά του. Τέτοιοι εργαζόμενοι είναι επιρρεπείς σε κακή ποιότητα ύπνου ή η κακή ποιότητα εργασίας αυξάνει τον την πιθανότητα να παραπονιέται κανείς για κόπωση. Σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες και τις διακριτική ευχαίρεια, περισσότερη αυτονομία αυξάνει την πιθανότητα να έχει καλύτερο κανείς ύπνο ή να μην υποφέρει από πονοκεφάλους. Τώρα, επανασυμφιλίωση ή καλύτερο συνδυασμό εργασία και προσωπική ζωή. 19% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι δεν μπορούν να συνδυάσουν καλά την εργασία και την προσωπική ζωή. 81% μόνο. Ε, έχουν θετική εμπειρία. Και οι άντρε περισσότερο ε, θεωρούν ότι είναι ο συνδυασμό πιο εύκολος, γιατί οι γυναίκες περισσότερο διαλέγουν εργασιακές ώρες ε, και ρυθμίσει εργασιακές ε, που συνάδουν με την προσωπική του ζωή. Αλλά οι γυναίκε έχουν και πολύ περισσότερε μη αμοιβόμενε εργασίε και λιγότερη ένταση εργασία έχουν όταν μένουν στο σπίτι για τα παιδιά. Οπότε αρνητικά συνδέεται ο συνδυασμό με τις μακρές και άτακτες ώρες εργασίας, ενώ θετικά με τις συντομότερε ώρες, την αυτονομία κτλ. Και η δυνατότητα επίση τηλεργασία, που συνάδει με το, με το συνδυασμό εργασία και προσωπική ζωή. Τώρα και εδώ έχουμε κάποιες, κάποιους δείκτες για την ποιότητα της εργασίας. Όσο πιο μεγάλη η ποιότητα της εργασίας, τόσο πιο εύκολος ο συνδυασμός εργασίας και προσωπικής ζωής. Και εδώ είναι αμφίδρομη η πορεία. Με θετικό τρόπο στο συνδυασμό και με αρνητικό τρόπο να συνεχίσει κανείς να να προβληματίζεται με τη δουλειά του, τότε δεν έχει χρόνο για το σπίτι, είναι πολύ κουρασμένος το φυσικό περιβάλλον επίση αυξάνει τη δυνατότητα να είναι κανεί υπερβολικά κουρασμένο μετά τη δουλειά. Το ίδιο ισχύει για την ένταση εργασία και αυτό αυξάνει την πιθανότητα να δηλώσει ο εργαζόμενο ότι συνεχίσει να προβληματίζεται για τη δουλειά του. Και επειδή ο χρόνο τρέχει, να περάσω στην επόμενη, στην επόμενη διαφάνεια. Ε, άνηση κατανομή τη μη αμοιβόμενη εργασία. Αυτό εξαρτάται φυσικά από την παρουσία των παιδιών στο νοικοκυριό. Ε, ενώ οι άνδρες που ασχολείται σε τέτοιε μη αμοιβόμενε εργασίε, δηλαδή οικιακέ ε, εργασίε και παροχή φροντίδα. Ο αριθμό των ανδρών αυξάνεται ιδιαίτερα όταν γίνονται παιδιά. Άρα είναι από 5 ώρες την εβδομάδα όταν δεν υπάρχουν παιδιά μέχρι 20 ώρες ε, όταν υπάρχουν παιδιά. 12 μέχρι 30 για τις γυναίκες όταν υπάρχουν παιδιά. Φυσικά μειώνεται αυτός ο αριθμός όταν, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά. Και επίσης ε, αυξάνεται για τις γυναίκες άνω των 60 που προς το τέλος ε, ε, του κύκλου εργασίας τους αυξάνεται η μη αμοιβόμενη δουλειά. Και τέλος, ε, είναι σημαντικό συνδυασμό εργασία και προσωπική ζωή και η ικανοποίηση των διαφόρων αναγκών μπορεί να γίνει σε διαφορετικά επίπεδα. Δεν υπάρχει μία νέα λύση για όλους. Πάντως, το όλο νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικό. Διαφορετικές ανάγκες υπάρχουν και μάλιστα, διαφορετικές λύσεις θα πρέπει να προκριθούν. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αντιμετώπιση, θα πρέπει να βρούμε ελαστικές ρυθμίσεις. Και μάλιστα μερικές λύσεις δεν χρειάζεται να είναι καν μόνιμες, μπορεί να είναι αναγκές μόνο προσωρινά. Ισότητα των δύο φύλων και Συνδυασμό εργασία και προσωπική ζωή. Πολύ σημαντικά θέματα, αν θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουν οι εργαζόμενοι να παραμένουν στην εργασία του μέχρι αργά, σε προχωρημένη ηλικία. Και φυσικά ισότητα δωρό και γυναικών. Και η ποιότητα εργασία ε, έχει σχέση με την βιωσιμότητα τη εργασία και τον συνδυασμό εργασία και προσωπική ζωή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχοντας ακούσει αυτή την παρουσίαση, καταλαβαίνουμε πόσο το Ίδρυμά σας έχει σημασία στην έρευνα κοινωνικών ζητημάτων. Ιδίως στην έρευνα των συνθήκων εργασίας στην Ευρώπη. Δεν θα καθυστερήσω για να έχουμε χρόνο για ερωτήσεις και συζήτηση μετά, να περάσω απευθείας στον επόμενο πανελίστ, μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κίστενσεν, ευχαριστώ. Είμαι, ήμουν εισηγητή για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Υγεία και την Ασφάλεια όταν έγινε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε περισσότερα για να έχουμε βιώσιμη εργασία. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σημαντικό είναι να έχουμε υψηλής ποιότητας τεκμηρίωση, όπως ακούσαμε, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορούμε όντως να αναλάβουμε δράση για τα σημαντικά ζητήματα. Επίσης, θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ε, κοινά νομικά πρότυπα για την εργασιακή ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τη σχετική της πρόταση και ελπίζουμε ότι το πλαίσιο που θα προτείνουν για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θα είναι φιλόδοξα το Δεκέμβριο. Δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν. Όμως και εμείς οι πολιτικοί έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε. μπορούμε να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποβάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο, διότι το πλαίσιο υγείας και ασφάλεια όπως προτάθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο, συγκέντρωσε συντριπτική πλειοψηφία, λέγοντας ότι το θέμα αυτό προέχει και για μας. Θεωρώ επίσης ότι οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες μπορούν να κάνουν πολλά από την πλευρά τους, λόγω του κοινωνικού διαλόγου που έχει θεσπιστεί. Από εκεί μπορεί να προκύψουν καλές προτάσεις. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στις υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Είμαι υπερήφανος γιατί προέρχομαι από μια χώρα όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να ζήσουν με το μισθό τους. Ό,τι και αν κάνουν έχουν αξιοπρεπή ζωή. Ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό και αν κοιτάξει κανείς ότι ένας στους πέντε δεν έχει ποιοτική θέση εργασία, δίκαια του μισθού και τι εργασιακέ συνθήκε, καταλαβαίνει πολλά. Εάν πρέπει να δουλέψει κανεί περισσότερε ώρε για να έχει ένα εισόδημα τη προκοπή, εάν πρέπει να πιάνει δεύτερη δουλειά για να έχει χρήματα να ζει στη ζωή του και την οικογένειά του, θα είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα και για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως με τις μειοκινητικές διαταραχές. Αν θέλουμε ο κόσμος να παραμένει περισσότερο στην αγορά εργασία, πρέπει να είναι και σε καλή υγεία. Πρέπει να έχει τη σωματική κατάσταση για να το κάνει αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που θα πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας. Εάν δείτε τι κάνουν οι διάφορες εταιρείες, οι εργοδότες, έχουν τη δυνατότητα θα θέλουν να κρατάνε τους εργαζομένους περισσότερο καιρό στη δουλειά τους. Δεν θα είναι εναντίον τους να είναι εξωπρεπέστερες συνθήκες εργασίες, ξέρουμε ότι από τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, υγεία και ασφάλειας το κόστο είναι τεράστιο για όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι θα μειώσει κανείς και το κόστος των κρατών μελών με περισσότερη υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Νομίζω σημαντικό είναι και από την οπτική γωνία των εργοδοτών, το λέω σοσιαλιστής, από την ε, οπτική γωνία λοιπόν των εργοδοτών να επικεντρωθούν στους εργαζομένους και να τους αντιμετωπίσουν ως πόρος, όχι ως κόστος. Οι εργαζόμενοι να μπορούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στην εργασία τους και να εξελιχθούν σε σταδιοδρομία τους σε μια εταιρεία κάνοντας διαφορετικά πράγματα. Πολύ σημαντικό για όλες τις χώρες να το σκεφτούν. Όμως αυτό απαιτεί Απαιτεί ανάπτυξη. Ένα φάσμα πρωτοβουλειών από του κοινωνικού εταίρου, από του πολιτικού ευθύνοντε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνουν οι κατάλληλε προτάσει. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ήθελα να σας κόψω στη μέση της πρότασή σας. Αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε περισσότερο χρόνο για το τέλος, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με το κοινό, γιατί ως τώρα τα έχουμε πάει καλά. Και τώρα να σας ε, παρουσιάσω την ε, Κρίστα. Κρίστα Σέντλατσεκ, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφαλή στην Εργασία. Γεια σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ευχαριστώ και τον κύριο Φάουντ για τη μελέτη και την έρευνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Φάουντ διότι ενημερωθήκαμε γέρο για τον αντίκτυπο και τα αριθμητικά στοιχεία τη μελέτη, και τώρα θα παρουσιάσουμε ένα νέο εργαλείο στον ιστοτοπό μα. ένα εργαλείο ε, που επιτρέπει να έχουμε εικόνα όλων αυτών των δεδομένων. Θα εξηγήσω γιατί το χρησιμοποιήσαμε και εκεί θα δούμε όλα τα δεδομένα και τους αριθμούς σαν μια χαρτογράφηση της Ευρώπης αλλά και όλου του κόσμου ε, για την διαχείριση και την γυράσκουσα εργατική δύναμη. Ε, θα είναι σημαντικό να εμπλουτίζουμε διαρκώς αυτά τα δεδομένα. Ίσως να εξηγήσω λίγο τι κάνουμε εμείς στον όσα στον οργανισμό μας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, για μια βιώσιμη εργασιακή ζωή. Ξέρουμε, ξέρετε ότι επικεντρωνόμαστε στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. χρόνο παραχρόνο οργανώνουμε μία διάσκεψη. Πέρσι οργανώσαμε κάτι για τους υγιείς εργασιακούς χώρους ασχέτως ηλικία. Τώρα είμαστε στον ενδιάμεσο χρόνο και κοιτάζουμε ήδη πόσο ενδιαφέρονται τα κράτη-μέλη σε επίπεδο σχεδιασμού πολιτική αλλά και εταιριών, αλλά και κοινωνικών εταίρων και κυβερνήσεων, πόσο θέλουν να πετύχουν περισσότερη ε, ενημέρωση και συγκέντρωση γνώσεων. Και κυρίω όλα αυτά κάποια στιγμή να φτάσουν και στο επίπεδο των εταιριών και επιχειρήσεων για να δουν ποια εργαλεία, ε, στρατηγικέ, πρακτικέ μπορούν να εφαρμοστούν. Το ιστορικό, τα θεμέλια για την εκστρατεία μα για τους υγιεί εργασιακούς χώρους ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει πιλωτικό πρόγραμμα για την ε, ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σχέτω ηλικία, αλλά με περισσότερη έμφαση στου πιο ηλικιωμένου εργαζομένου. Τι κάνουμε. Αναλύουμε την κατάσταση όλων των κρατών μελών, ακόμα και εκτός της Ευρώπης, με τις υπάρχουσες πολιτικές πρωτοβουλίες για να αντιμετωπιστεί η γύρανση του εργασιακού πληθυσμού. Και κοιτάζουμε πώς εφαρμόστηκαν οι διάφορες πρωτοβουλίες στα κάτι μέλη και εκτός στις υπόλοιπες χώρε μέλη. Ε, έπειτα θέλαμε να έχουμε ένα σύνολο βιώσιμων πληροφοριών και αναλυτικών στοιχείων για τις πολιτικές επιλογές με, την, ε, με στόχο την, την αποκατάσταση και την επιστροφή στο χώρο εργασία, ακόμη και σε εθνικό, περιφερειακό, τομεακό επίπεδο. Τέλος, θέλαμε ανταλλαγή καλών πρακτικών σε επίπεδο χωρών. Αυτό ήταν το σημείο αφετηρίας, ο στόχος. Τώρα, βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε δημοσιεύσει στον ιστότοπό μα εκθέσει για 28 κρατημέλη. Βλέπουμε τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Επίση έχουμε πολλά case studies, μελέτε ειδικών περιπτώσεων, με ανάλυση για να δούμε πώ μπορούν να αξιοποιηθούν όλα αυτά σε επίπεδο εταιρεών και επιχειρήσεων και έχουμε και στοιχεία για την αποκατάσταση και την επιστροφή στον χώρο εργασία. Επίση, μια παρατήρηση γιατί ταιριάζει με αυτά που ακούσαμε προηγουμένω. για τα στοιχεία, τους αριθμούς και την ποιότητα στην ε, εργασία. Ιδίω για το δομικό πλαίσιο και για να πετύχουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Όπως προείπα, χαρτογράφηση των εθνικών στρατηγικών και πολιτικών και να αναφέρω απλώς κάποια στοιχεία επιτυχών πολιτικών επιλογών. Εδώ υπάρχει και ένας στενός συσχετισμός με την ποιότητα της εργασίας. Οι πλέον επιτυχείς χώρες, και πρέπει να πω ότι είναι μετρημένες στα δάχτυλα, είναι πολύ επιτυχημένες στον τομέα αυτό. Γιατί? Γιατί μπόρεσαν να έχουν μια προσέγγιση σφαιρική, προσέγγιση ομπρέλα. Μπόρεσαν να ενσωματώσουν διαφορετικές πολιτικές επιλογές στο πλαίσιο τους με μίζο στόχο να διατηρήσουν την απασχολησιμότητα και την εργασιμότητα όλων των εργαζομένων. Εδώ μιλάμε για απασχόληση, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, δημόσια ασφάλεια και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχει κεντρικό συντονισμός με χρηματοδότηση, κοινωνικό διάλογο, πολύ σημαντικό αν θέλουμε να πετύχουμε. Ένα μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε, διότι ξέρουμε ότι όλα τα κρατη μιλη αυξάνουν το όριο συνταξιοδότηση, μπορούμε να πούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσει στα συνταξιοδοτικά χωρί ανάλογε πολιτικέ για να ε, διατηρηθεί η αποσχολησιμότητα μέσω τη δυνατότητα απασχόληση, δηλαδή εργασιμότητα όλων των εργαζομένων και την συμμετοχή σημαντικών κοινωνικών εταίρων με κοινωνικό διάλογο και την υιοθέτηση την, ε, μιας ε, διαβίου επαγγελματικής ε, προοπτικής. Μόνο έτσι θα πετύχουμε και τα πορίσματα αυτά τα δέκα στον ιστοτοπό μας. Το ίδιο και για την αποκατάσταση και την επιστροφή στα εργασιακά συστήματα. Παρόμοια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν περισσότερα απομετρημένα στα δάχτυλα τα κράτη-μέλη που είναι πολύ πετυχημένα, οπότε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση και για του υπόλοιπου. Και εδώ θα πρέπει να συνδυάσουμε πολιτικά και νομικά πλαίσια με συμμετοχικά συστήματα, με έγκαιρη παρέμβαση, ιδίως σε επίπεδο εταιρεία επιχείρησης, ε, μια ε, στοχευμένη, σχεδιασμένη ειδικά για το κάθε πρόσωπο, για το κάθε άτομο, ώστε να καλύπτω οι ανάγκε του προσέγγιση και μηχανισμού συντονισμού. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο ή τομεακό ή ασφαλιστικό, αλλά και σε επίπεδο εταιρεία επιχείρηση. Αυτά κοιτάμε στα συστήματα αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία. Τώρα το πλέον σημαντικό για μα, για την εκστρατεία μα για του υγιεί εργασιακού χώρου, είναι να κοιτάξουμε τι είναι σημαντικό για τι επιχειρήσει, τι εταιρείε, του εργοδότε, του εργαζομένου, του κοινωνικού εταίρου. Τι είναι σημαντικό να βελτιωθεί. Ω προ την εργασιμότητα, δηλαδή την δυνατότητα απασχόληση σε επίπεδο εταιρεία. Βλέπουμε μία ε, προσέγγιση του βίου, του επαγγελματικού βίου. Εδώ μιλάμε για όλους τους εργαζομένους. Μιλάμε για μια ε, διαδικασία που να ξεκινήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα, με παρέμβαση σε επίπεδο εταιρεία επιχείρηση. Επίση, ακούσαμε ήδη σήμερα ότι μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε εδώ μελέτε αντικτύπου, δηλαδή διαφορετικέ πολυφωνικέ μελέτε αντικτύπου, ώστε να ε, μελετηθούν όλοι οι κίνδυνοι με τα προβλήματα στον χώρο εργασία, τα κοινωνικά προβλήματα, στενή συνεργασία μεταξύ των ανθρωπίνων πόρων και το, του μάνατζερ για την υγεία και την ασφάλεια. Αναφέρθηκε ο ηγετικό ρόλο που πρέπει να αναλυφθεί, δηλαδή για να έχουμε καλύτερη ποιότητα και εργασιακέ συνθήκε. Η ε, ανάληψη ηγετικού ρόλου είναι πάντοτε σημαντική και μετά ο κοινωνικό διάλογο και η συμμετοχή των εργαζομένων. Αυτά ήταν η βάση και τα θεμέλια. Έρχομαι στα τελευταία σχόλια. Αυτή ήταν η βάση για την εκστρατεία για τους υγιείς χώρους εργασίας. Μήνυμα που ε, απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα, όμως ε, εν τέλει πρέπει να συναντηθούμε με τους υπευθύνου των εταιρεών και των επιχειρήσεων ώστε να προβλεφθούν αλλαγές αφού συζητηθούν με όλους τους εταίρους. Όλους τους ενδιαφερομένους συνομιλητές. Αυτή η εκστρατεία λοιπόν είχε τρεις μέγιστους στόχους. Πρώτον, να προωθήσουμε τη βιώσιμη εργασία, προ παρέχοντας τις πληροφορίες που διαθέτουμε ήδη με συγκεκριμένα στοιχεία και αριθμητικά δεδομένα, έπειτα ιδιαίτερη σημασία πρόληψης και παρέμβασης καθόλου τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, να μην ξεκινήσουμε με τη γενιά των 45 συν και μετά η στήριξη των εργοδοτών και εργαζομένων με την παροχή πληροφοριών και εργαλείων. Υπάρχουν εργαλεία, υπάρχουν στρατηγικές και προγράμματα, ε, τα παρουσιάζουμε ήδη στις εταιρείε και τι επιχειρήσει, ακόμα και στι μικρομεσαίες, Οπότε μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά μπορούν να επιληθούν, αλλά πρέπει να καταπληθούν προσπάθειες. Όπως πάντοτε στις εταιρείε και τις επιχειρήσεις, στήριξη χρειάζεται από τους μάνατζερ, από τη δίκηση. Ε, και πρέπει να ξεκινήσει από ψηλά η διευκόλυνση όλης αυτής της διαδικασίας. Αυτά από πλευρά μας ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ και βλέπουμε εδώ ακριβώς την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ του ταμείου σα ε, και τον λοιπόν. Ένα σχόλιο λοιπόν το οποίο ε, έκανα για αυτά τα ενδιαφέροντα που είπατε είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει αλλαγή των ε, συνταξιδοτικών συστημάτων χωρίς να εξετάζουμε την απασχολησιμότητα των ηλικιωμένων εργαζομένων. Τώρα να παρουσιάσω άλλο έναν συνάδελφο από τα θέματα των κοινωνικών και της απασχόλησης την Τατιάνα, πράσινη και διακεκριμένο μέλος της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Μαριάν και ευχαριστώ και το Φαν... Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που παρουσίασαν αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Πρέπει βεβαίως να δούμε τα πράγματα εις βάθος, αλλά αρκετές πληροφορίες παρόλα αυτά. Οπότε, εγώ βρίσκομαι εδώ, λόγω της έκθεσης που εγκρίναμε το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια για την δημιουργία συνθήκων στην αγορά εργασίας που θα ευνοούν την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Ήταν μια έκθεση από δύο επιτροπές, Επιτροπή Απασχόλησης και Γυναικών, με δύο συνεισηγήτριες, την κυρία ναι, Τε. Ε, αλλάζουν τα, τα ονόματα εκεί στα λιθουανικά ανάλογα με το αν δεν ξέρω, με την κατάσταση της γυναίκας. Και η άλλη συνεισηγήτρια ήμουν εγώ. Από κέντρο αριστερά, σοσιαλιστές και πράσινοι και από δύο χώρες, ε, Λετωνία και Λιθωνία. Υπήρχε όμως στήριξη παρόλα αυτά για την τελική έκθεση. Μία ομάδα, οι συντηρητικοί, καταψήφισαν το Κοινοβούλιο κυρίως ε, στήριξε. Τα υπόλοιπα τμήματα του Κοινοβουλίου στήριξαν την έκθεση. Και βεβαίω. Σημασία έχει η ιδιωτική ζωή και, και Βεβαίω ε, και η εργασιακή ζωή και η οικογενειακή ζωή. Και βεβαίω έχουμε, ακούσαμε και τα ευρήματα της έρευνας. Η δικιά μας η θέση όμως σε γενικές γραμμές συμπίπτει με τα ευρήματά σας και βεβαίως εδώ πέρα αυτό το οποίο κάνει δύσκολη την κατάσταση, αλλά και εύκολη ίσως είναι ότι δεν υπάρχει μια ενιαία λύση για όλους. Δηλαδή, η λύση για να συνδυαστεί η οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες σε διαφορετικές χώρες, περιφέρειες και οικογένειες. Αυτό το οποίο λέγαν παλιά ήταν 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση και 8 ώρες διασκέδαση. Ε, βεβαίω δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα τώρα. Η κατάσταση αλλάζει. Υπάρχει βεβαίω ε, και η διαδρομή που κάνει κανείς να πάει στη δουλειά του και οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την τηλεεργασία. που ε, βεβαίως σημαίνει και περισσότερη ευελιξία. Επίσης στην έκθεσή μας κάνουμε προτάσεις μη νομοθετικές αλλά και νομοθετικού χαρακτήρα ε, που είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο προτείναμε στην έκθεσή μας πρώτα απ' όλα είναι ε, οι οικογένειες με παιδιά όπου βλέπουμε ακόμα μεγάλα κενά χάσματα στις ευθύνες ανδρών και γυναικών. βεβαίως ε, δεν πρέπει να επηρεάζεται η απόφαση των οικογενειών να κάνουν παιδιά από το εισόδημα. Και δεν πρέπει βεβαίως να υποβιβάζει το επίπεδο ζωής. Και δεν υπάρχει ακόμα ισχυρή νομοθετική βάση για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, προτείνουμε σε όλα τα κράτη-μέλη, στους κοινωνικούς εταίρους, να ξαναδούν το σύστημα αποζημίωσης για την γονική άδεια για να υπάρχει μια αντικατάσταση του εισοδήματο που θα είναι επαρκής και βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχει και γονική άδεια μετά από τα νόμιμα την ελάχιστη εγγυημένη περίοδο. Βεβαίω υπάρχει μια μεγάλη ε, συζήτηση για την ε, ε, γονική άδεια που μεταφέρεται και αυτή που δεν μεταφέρεται. Κάποιοι εκπρόσωποι ειδικά αριστερών ομάδων ζήτησαν να μην ε, μεταφέρεται η γονική άδεια, αλλά η συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων ήταν ότι μεγάλο κομμάτι πρέπει να μην μεταφέρεται, αλλά να υπάρχει μια ευελιξία. Και επίσης η γονική άδεια μπορεί να ξεπεράσει και το ελάχιστο νόμιμο διάστημα και βεβαίως ε, την ηλικία του παιδιού και η θέση μας είναι ότι πρέπει να υπάρχει ισότητα των δύο γονιών και οι δύο γονείς βεβαίως να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το οποίο προτείνουμε λοιπόν ως νομοθετικό μέσο. Είναι σημαντικό η Κομισιόν να προτείνει πρωτοβουλίες όπως οι αδιαπατρότητες. Με κάποιο ελάχιστο βεβαίω. Δύο εβδομάδες ε, πληρωμένης άδειας υποχρεωτικές. Μια άλλη οδηγία που θέλουμε να συζητήσουμε με την Κομισιόν είναι η οδηγία για την άδεια των ατόμων που φροντίζουν άλλα άτομα. Ξέρετε πως ε, τον καιρό μας ο χρόνος που αφιερώνεται σε φροντίδα ε, συνεχώς αυξάνεται. και δεν είναι θέμα φροντίδας ε, παιδιών μόνο, αλλά και ηλικιωμένων και άλλων ε, μελών της οικογένειας. Προτείνουμε λοιπόν να υπάρξουν κάποιες πιστώσεις ε, για την φροντίδα ατόμων μέσω της νομοθεσίας και για άντρες και για γυναίκες. και βεβαίω αναθεμελιώνονται και συνταξιδοτικά δικαιώματα για όσους διακόπτουν την ε, σταδιοδρομία τους για να φροντίσουν ε, κάποιο μέλος οικογένειας ή κάποιον άλλον. Και βεβαίως Ε, και σε αυτή την οδηγία θα πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι οι άνδρες και οι γυναίκες και να ε, χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες ε, και από τους δύο. Αν το επιβάλλουν οι οικογενειακές συνθήκες. Οπότε, αν έχετε άλλες ερωτήσεις, ευχαριστώ να ε, απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε, Τατιάνα. Ανέφερε την υποστήριξη που δέχτηκες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτό δείχνει την ποιότητα της έκθεσης. Γι' αυτό και υποστηρίχθηκε τόσο ενθουσιοδός. Τελευταίος ο μιλητής από το πάνελ αυτό είναι ο Γιώχαν. Είπα να μην επιχειρήσω να, να προφέρω το ε, επιθετό σου. Είναι από τη Γενική Διεύθυνση ε, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Καταναλωτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Είμαι ο τελευταίος ομιλητής αυτού του πάνελ και είχα κάποιες ιδέες για το περιεχόμενο της ομιλίας μου, αλλά ενδόμηχα ελπίζα να με προκαλέσουν οι προλαλήσαντες με κάποιες ε, αμφιλεγόμενες ιδέες τους, οι επίμαχες. Αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν άκουσα τίποτα ε, που να ε, να προκαλεί τη διαφωνία. Οπότε, για να έχουμε και μια ζωηρή συζήτηση, θα ήθελα να σας παραπέμψω στα πορίσματα της έκτης έρευνας, επισκόπησης για τις εργασιακές συνθήκες του Ιδρύματος Eurofound και να σας αναφέρω τα βασικά σχέδια που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην οδηγία για την, στην Γενική Διεύθυνση ε, Ισότητας αλλά και στην Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης στην οποία απασχολούμαι εγώ. Χωρίς όμως να επισέρχομαι σε υπερβολικές λεπτομέρειες. Για τη δική μας διεύθυνση εξετάζουμε τα σημεία που αφορούν ιδιαίτερα το συνδυασμό εργασίας και προσωπικής ζωής. Βέβαια, δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω από τώρα το περιεχόμενο της ανακοίνωσης ε, που πρόκειται ε, όσον ούπο να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ασχοληθώ με τις πτυχές εκείνες που έχουν σχέση με το δικό μας έργο της προσπάθειας καταπολέμησης των διακρίσεων ε, μεταξύ των δύο φύλων. Γιατί υπάρχουν εκεί πολλά κοινά σημεία Επίσης, ε, προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τις διακρίσεις λόγω ηλικίας, αλλά εξετάζουμε και τη θέση των ε, πιο ηλικιωμένων εργαζομένων και των ηλικιωμένων γενικώ. Ε, θέματα που ρητά ανέφερα και μερικοί προλαλήσαντες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πορίσματα της επισκόπησης του Eurofound, θα ήθελα να σταθώ σε μερικά πορίσματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα για τη χάραξη των δικών μας πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σας ε, εκφράσω επ' και κάποιες ευχές μας. Γιατί είμαι βέβαιος ότι ήδη στο βιβλίο αρχίσατε να ε, εξετάζετε, να σκέφτεστε από τώρα την 7η επισκόπηση. Μπορεί να είναι λίγο νωρίς, αλλά ποτέ δεν είναι ε, αρκετά νωρίς για τέτοιες σκέψεις. Κάποια ενδιαφέροντα πορίσματα της επισκόπησης. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη γύρανση του εργατικού δυναμικού. Το 2005, 24% του εργατικού δυναμικού ήταν άνω των 50 ετών. Δέκα χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, το 2015, ήδη τριδέν είναι το ποσοστό των εργαζομένων άνω των 50. Κάτι που θα έχει σημαντικές ε, συνέπειες ή επιπτώσεις και στη ζήτηση της ποιότητας της εργασίας. Και δείχνει επίση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ε, σχετικά επιτυχής στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των εργαζομένων. Βλέπετε από τα στατιστικά στοιχεία ότι κάθε χρόνο αυξάνεται αυτό το ποσοστό απασχόλησης και πιστεύω ότι αυτή η ανωδική πορεία θα συνεχιστεί. Που σημαίνει ότι η παροχή των σωστών θέσεων απασχόλησης για τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Ε, Εξέτασε και κάποια πορίσματα που αφορούν τη διάκριση των φύλων Υπάρχει δυστυχώς θέμα διακριτικής μεταχείρισης. Και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των φύλων σε ό,τι αφορά τις παραμέτρους ποιότητας των θέσεων εργασίας. Γενικώ η κατάσταση βέβαια δεν είναι δραματική, ιδιαίτερα απογοητευτική, οπότε κατά τη γνώμη υπάρχει κάποια εξισορρόπηση. Πάντως η διαφορά μεταξύ των φύλων ε, επιβεβαιώνεται και από την μελέτη της Eurofound και απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τώρα τη βιώσιμη απασχόληση. Το εξετάζουμε υπό το φως της ψηφιοποίησης, της ρομποτοποίησης ε, των θέσεων εργασίας και στη μελέτη της Eurofound, του Eurofound ε, δίνεται μία μερική μόνο απάντηση σε πολλές ερωτήσεις. Ο ενδιαφέρον δείκτης από την άποψη αυτή είναι ο δείκτης για την ποιότητα του ωραρίου εργασίας. Και πάλι βλέπουμε διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά δεν είναι τόσο εντυπωσιακέ. Παρόλο που και εδώ υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των φύλων. Αλλά το χάσμα δεν είναι τόσο μεγάλο και είναι ενδιαφέρον αυτό. Από τη μια έχουμε μεγάλη διαφορά στις, ε, στο διαχωρισμό των θέσεων εργασία, αλλά σε ό,τι αφορά την ε, ποιότητα δεν υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Το ίδιο ισχύει και τους άλλους δείκτες. Ε, το πόσο τακτικέ είναι οι ώρε εργασία, εδώ είναι σε καλύτερη θέση οι γυναίκες που έχουν πιο τακτικά ωράρια. Και ένα άλλο δείκτη που εξέτασα και που αφορά σε κάποιο βαθμό τις δικές μας προσπάθειες για καταπολέμηση των διακρίσεων, ο δείκτης για το κοινωνικό περιβάλλον. Σας τον συστήνω. Απαρτίζεται από 15 επιμέρους δείκτες και δύο υποκατηγορίες. Την ε, συνέπεια της ε, δυσμενούς ε, κοινωνικής συμπεριφοράς ή το αντίθετο η εμφάνιση υποστήριξης. Είναι πολύ σημαντικά στοιχεία που επηρεάζουν ε, τον δίκτυο αυτό του κοινωνικού περιβάλλοντος και μας εμπνέουν ε, για τις πολιτικές που θα ακολουθήσουμε στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά την προοπτική των φύλων, μια άλλη ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι το στοιχείο για τις γυναίκες σε θέση μάνατζερ. Βέβαια, ακόμη έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε, αλλά έχουμε και ένα σχετικά θαρρυντικό πόρισμα τον αριθμό των γυναικών σε θέση μάνατζερ που έχει αυξηθεί. Επίσης, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν γυναίκες προϊσταμένους. Αυξάνεται ο αριθμός αυτός. Και μάλιστα η πλειοψηφία και των γυναικών εργαζομένων έχει γυναίκα προϊσταμένη. Και βέβαια αυτό σχετίζεται με τις διαφορές τη ε, της παρουσίας των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, αλλά παρόλα αυτά η αύξηση των ε, ε, γυναικών σε ηγετικέ θέσεις είναι ενθαρρυντικό στοιχείο. Έχουμε πολλά στοιχεία που αφορούν τις διακρίσεις των δύο φύλων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη δυσμενή κοινωνική συμπεριφορά ή κάποια άμεσα ευρήματα για τις διακρίσεις. Με προβληματίζουν κάποια ποσοστά, γιατί θεωρώ ότι είναι λυπής η ενημέρωση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διάκριση λόγω ηλικία ή λόγω φύλου. Γιατί ε, δεν είναι πολλοί οι εργαζόμενοι που καταγγέλουν τέτοιες διακρίσεις. Γι' αυτό υπάρχουν λυπή στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τις διακρίσεις λόγω εθνοτικής καταγωγής, φυλής, ε, χρώματος, ε, δέρματος ή εθνικότητα. Είναι χαμηλά τα ποσοστά, 1 με 3%. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ χαμηλά έχουμε αμφιβολίες για το κατά πόσο γίνονται οι καταγγελίες όταν υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις. Κάτι που βεβαιώνεται και αυτό ε, σε πολλά πορίσματα της επισκόπησης του Ευρωβαρομέτρου είναι ότι η διάκριση λόγω ηλικία ε, είναι η εμφανέστερη μορφή διάκρισης στον χώρο εργασίας και θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να ξεχωρίσω ιδιαίτερος και να σταθώ σε αυτό στην απογευματινή συζήτηση, αφορά τον αυξανόμενο, την αυξανόμενη αναλογία ε, πιο ηλικιωμένων ε, εργαζομένων και τι πρέπει να κάνουμε για να τους κρατήσουμε όσο το περισσότερο χρόνο στην εργασία τους. Θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, λογικές ρυθμίσεις για να τους ικανοποιήσουμε. Τέτοιου είδους συλλογικές ρυθμίσεις ε, προβλέπεται στην οδηγία του 2000, 2078 που προβλέπεται χρέος ε, του εργοδότη να προσφέρει κάποιες συλλογικές ρυθμίσεις ε, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος έχει αναπηρήσει. Για το στοιχείο αυτό υπάρχει υποχρέωση, αλλά δεν ισχύει αντίστοιχη υποχρέωση να ικανοποιηθούν με λογικές ρυθμίσεις και άλλοι εργαζόμενοι, για παράδειγμα πιο ηλικιωμένοι, ενώ υπάρχει αυτή η ανάγκη. Και αναφέρθηκε το 1 τρίτο των εργαζομένων ε, λέει, αναφέρει ότι επωφελείται από τέτοιου είδους ε, ε, λογικές ρυθμίσεις παρόλο που δεν αποκαλούνται έτσι. Αλλά είναι μειοψηφία των εργαζομένων που ικανοποιούνται από τέτοιου είδου διευθετήσει. Φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ζητούν τέτοιε διευθετήσει, ιδιαίτερα στο μέτρο που προχωρούν στην ηλικία. Γι' αυτό και αντίστοιχη υποχρέωση ε, που υπάρχει για τους ε, εργαζόμενους με αναπηρία θα πρέπει να επεκταθεί και στους υπόλοιπους εργαζομένους. Και πριν από ένα χρόνο είχαμε μια μελέτη για τέτοιου είδου. Ε, ε, λογικές διευθετήσεις για τους εργαζομένους με αναπηρίες στον χώρο εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νομική μεταχείριση του θέματος αυτού στα κράτη-μέλη. Αλλά επαναλαμβάνω, επικεντρώμαστε μόνο στα άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να διευρύνουμε ώστε να προσφέρονται τι δυνατότητε λογικών διαθετήσεων και σε άλλε κατηγορίε εργαζομένων. Αυτά και μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Thank you very much, Johan. And I think you have given us some... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω πως αυτό το οποίο είπες ειδικά τελευταία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε 25 λεπτά ακόμα και δύο σχολιαστές. και η οποία είναι αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου της Αγοράς Εργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Βλαδιμίρα, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε και την δυνατότητα να μιλήσω κι εγώ στο πάνελ για την ε, έρευνα αυτή. Βεβαίως η έρευνα ήταν εμπιστευτική, αλλά πολλά νούμερα ήδη κυκλοφορούν. Εγώ εκπροσωπώ τους εργοδότες ε, και ευρύτερα θα έλεγα τους κοινωνικούς εταίρους και πολλές φορές στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οπότε γνωρίζω ότι η γύρανση των εργαζομένων είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να βρεθεί ένα καινοτόμο τρόπος προσέγγισης του κύκλου ζωή. Αναφέρθηκε και από την Κρίστα και από τον Όλεο ρόλο των κοινωνικών εταίρων και αυτός είναι ο λόγο για τον οποίο οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται μια αυτόνομη συμφωνία για την γύρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και μια τέτοια προσέγγιση το να λέμε απλά ότι οι εταιρείε χρειάζονται ανθρώπους όλων των ηλικιών, ότι πρέπει να είναι εργαζόμενοι υγιείς ε, και με προσόντα και δραστήριοι, ε, το υγιής βεβαίως αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας, τα προσόντα σημαίνει διαβίωση και δραστήριοι σημαίνει την δυνατότητα να παραμείνουν όσο θέλουν στην αγορά εργασία και βέβαια να ε, εμπλέκονται σε αυτό που κάνουν. Και βεβαίως αναφέρθηκε πως 89% ε, των ανθρώπων είναι ικανοποιημένοι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί τη μισή μας ζωή την περνάμε στη δουλειά. Και βεβαίως ε, πρέπει να το δούμε και από τη σκοπιά του ατόμου που εργάζεται και γυράσκει στον χώρο εργασίας και βεβαίως έχει διαφορετικές απαιτήσει ε, σε κάθε φάση για την ισορροπία ε, ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής. Υπάρχουν τρεις λέξεις που ακούγονται συχνά, η ευελιξία, η κινητικότητα και η ασφαλεία. Η ευελιξία αφορά η ασφάλεια αμφισβητείται συχνά. και βεβαίω ε, αφορά την ασφάλεια στη δουλειά αλλά και την δυνατότητα κανείς να απασχολείται. Θα πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι να έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν ε, τη ζωή τους ε, και την εργασιακή ζωή τους. Για τις ώρες εργασίας. Ε, δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα. 55% των ατόμων λένε ότι είναι ικανοποιημένοι από το ωράριο εργασίας ε, αυτή τη στιγμή. Και έρχομαι έτσι στην ισορροπία της επαγγελματικής με την προσωπική ζωή. Είναι πάρα πολύ θετικό το, το 81% των όσων απάντησαν θεωρούν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή ισορροπία. Οι άντρες είναι πιο θετικοί, αλλά από την άλλη οι γυναίκες... Οι άντρες είναι αρνητικοί, οι γυναίκες είναι πιο θετικές. Και βεβαίως μπορούν ε, να οργανώνουν καλύτερα και τα του νοικοκυριού και της ιδιωτικής ζωής. Και βεβαίως επειδή ο χρόνος περνάει γρήγορα. Δύο πράγματα στο τέλος για την συζήτηση. Επειδή η φύση της δουλειάς αλλάζει, οι άνθρωποι θέλουν να είναι πιο αυτόνομοι, να έχουν περισσότερο έλεγχο στη δουλειά τους, να κάνουν τη δουλειά τους όπως θέλουν και ιδιαίτερα η νέα γενιά της χιλιετίας, της νέας χιλιετίας δεν μιλάει για μια τέτοια προσέγγιση. Ε, οπότε δεν, δεν το βλέπουν ως πρόβλημα αυτή την ισορροπία εργασιακού και ιδιωτικού βίου. Και τέλος, ε, το θέμα της ρύθμισης. Αυτό το οποίο είπε η Τατιάνα, η πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν τόσες πολλές αλλαγές στην αγορά εργασίας που πρέπει να καταλήξουμε σε μια ρυθμισή στο επίπεδο της εταιρείας ε, μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Ε, δεν ξέρω δηλαδή αν απαιτείται περισσότερη ε, ρύθμιση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Βλαδιμίρα. Έκανες ένα σχόλιο προς την Τατιάνα ανέφερες και την ευελιξία και την ασφάλεια. Νομίζω πως όλοι έχει να πει δυο λογάκια, ίσως επ' αυτού. Ευχαριστώ και πάλι. Οπότε, ο τελευταίος σχολιαστής είναι ο Πάλο Παντσέρη, ο οποίος είναι στην Κόφασε για την ε, πολιτική και το login. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το Eurofund που μας κάλεσε σήμερα εδώ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό και τα αποτελέσματα της έρευνας. Θα αναφερθώ σε κάποια πραγματάκια. Να σας πω ποιοι είμαστε πρώτα απ' όλα. Η Κόφασε ιδρύθηκε το 1958. Έχουμε 59 μέλη σε 33 ε, χώρες και εκπροσωπούν γύρω στα 95 εκατομμύρια οικογένειες. Το θέμα λοιπόν αυτό μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και θα έλεγα ότι μαζί με άλλες ΜΚΟ που βρίσκονται εδώ πέρα σήμερα δημοσιεύσαμε ένα έγγραφο που λέγεται το Ευρωπαϊκό Πακέτο Συμφιλίωσης ε, Οικογενειακής και επαγγελματική ζωή, για να πούμε το τι σημαίνει αυτό για εμάς και είδαμε όλου τους τομείς που θεωρήσαμε σημαντικούς. Είχαμε ένα κομμάτι για άτομα που φροντίζουν, για τις υπηρεσίες ε, σε παιδιά, για την απασχόληση των γυναικών και τις λύσεις ε, στον χώρο εργασία. Και ένα θέμα το οποίο φροντίσαμε να προκύψει είναι ακριβώς η προσέγγιση του κύκλου ζωής, σε ολόκληρη τη ζωή. Γιατί τι σημαίνει για εμάς η συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι ότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε είναι ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα, δεν είναι επίδομα για τους νέους γονείς, δεν είναι κάτι για όσους δουλεύουν μόνο σε γραφεία είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να ισχύει για όλους τους εργαζόμενους. Ένας νέος τρόπος να δούμε την αγορά εργασίας, την οικονομία και την κοινωνία. Και επίσης πρέπει να δούμε και τις σχετικές πολιτικές και την ομοθεσία ως ένα δίκτυ ασφαλείας που υπάρχει ως διαφορετικά κομμάτια ενός παζλ που αποτελεί δηλαδή ένα δίκτυο ασφαλείας για τις οικογένειες που έχουν διαφορετικές ανάγκες σε κάθε στιγμή της ζωής τους. Οι οικογένειες δεν είναι κάτι το στατικό. Είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται, έχει και αυτό έναν κύκλο ζωής και υπάρχουν διάφορες οικογένειες. Κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές ανάγκες. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, διεθνείς οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες η λεγόμενη γενιά σάντουιτς που φροντίζει και τους γονείς και τα παιδιά της. Και πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο θα στηρίζει όλους αυτούς τους άνδρες και γυναίκες ε, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Της ζωής τους. Σύμφωνο λοιπόν με το ψήφισμα που λέω δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους. Και βεβαίω το πακέτο τη Κομισιόν που θα έρθει του επόμενου μήνε πρέπει να είναι φιλόδοξο, πρέπει να περιέχει νομοθετικά και μη νομοθετικά μέσα, και θα μιλάμε για νομοθετικά μέσα. Παραδείγματο χάρη ναι, εδώ πέρα σκεφτόμαστε κάποιο σύστημα αδεία, να έχουμε πληρέστερα πακέτα άδεια, μητρότητα, πατρότητα, γονική, για άτομα που φροντίζουν άλλους, ανεξαρτήτως του καθεστώτος απασχόλησης, αυτοαπασχολόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι έχουν παιδιά και έχουν ευθύνες να φροντίζουν άλλους. Και έρχομαι εδώ πέρα σε δύο πράγματα, σε κάποια πράγματα που θα ήθελα να δείξω. Υπάρχει αυξηνόμενη ανάγκη οργάνωσης, υπάρχει επισφάλεια, υπάρχουν δουλειές τις οποίες είναι κανείς ανα πάσα στιγμή στη διάθεση του εργοδότη. Δηλαδή η αυτοαπασχόληση είναι πάρα πολύ καλή αν το επιλέγει κανείς. Δεν μπορούμε όμως να πιέσουμε ε, προς αυτή την κατανησία να λέμε ότι αυτή είναι η μόνη λύση. Βλέπουμε ότι 20% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λένε ότι ο μόνος τρόπος που είχαν να βρουν δουλειά ήταν ε, ως αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, ε, Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα παιδιά, ή ε, τα παιδιά του ηλικιωμένου, ε, τα άτομα με αναπηρία. Αν δεν υπάρχουν υπηρεσίε για όλους αυτούς, τα αναλαμβάνει η οικογένεια. Και τι λέμε οικογένεια, συνήθως τι γυναίκες. Και δεν μπορούμε εκεί πέρα να μετρήσουμε συνθήκες εργασίας ε, ή ικανοποίηση για δουλειά, γιατί φεύγουν από την αγορά εργασία. Δεν είναι πια εργαζόμενοι. Ή υπάρχει σε μια τέλεια, φταία λύση, μερική απασχόληση. Εντάξει, καλή η μερική απασχόληση, δεν είμαστε εναντίον, αλλά αρκεί ο κόσμος να το θέλει. Όχι όταν είναι η μόνη λύση. Θεωρούμε λοιπόν πως υπάρχουν ε, και άλλοι ευέλικτοι τρόποι για να στηριχθούν οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι, να μην ε, πέσουμε σε μερική απασχόληση χαμηλής ποιότητας Επίσης ε, θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση με τους εργοδότες ε, για να υπάρχει μια ευελιξία στο ωράριο χωρίς να υποφέρει κανείς. Το είχαμε συζητήσει και το θέμα της ψηφιοποίησης στο Βερολίνο πριν από λίγες εβδομάδες. Η έξυπνη εργασία πρότεινε και το Κοινοβούλιο εδώ κάποια πράγματα. Ε, η τηλεεργασία 2,0 δηλαδή, το επόμενο βήμα. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν οι ψηφιακές ε, τεχνολογίες να μην οδηγήσουν ε, στο να μην είναι κανείς παρόν στη δουλειά, αλλά να είναι τελικά διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο μέσω email ε, και τηλεφώνου. Πώς ακριβώς θα βρεθεί αυτή η ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, να μην γίνονται όλα μια σούπα χωρίς μια διαχωριστική γραμμή. Και εδώ πέρα ίσως διαφέρει η άποψή μου λίγο από την προλαλή σας. Εμείς χαιρόμαστε που κάποιες εταιρείες προτείνουν ε, κάποιες ε, τέτοιες ε, εμπειρίες και θεωρούν πως οι κοινωνικοί εταιροί προσφέρουν διάφορες ευκαιρίες και οι εταιρείε έχουν σημαντική εμπειρία να μοιραστούν, αλλά θεωρούμε ότι ένα πλαίσιο το οποίο θα προστατεύει τους εργαζόμενους ε, και τους πιο ευπαθείς εργαζόμενους ειδικά είναι κάτι το πάρα πολύ χρήσιμο. Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας αυτό και θα ήθελα να πω πως πρέπει να υπάρχουν μέτρα νομοθετικά και μη νομοθετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Paolo, for that. Ευχαριστούμε Πάολα για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Έχουμε 10 λεπτά διότι θα ήθελα να κλείσουμε στην ώρα μας και θα χρησιμοποιήσω τα προνόμια της Προέδρου, διότι όλα όντω έκοψα λίγο νωρίτερα. Θα σου δώσω απλώς λοιπόν δύο επιπλέον λεπτά, ώστε να μπορέσεις να σχολιάσεις ό,τι θες από αυτά που άκουσες και μετά ο λόγος του κοινού μας. Σε ευχαριστώ πολύ Μαριαν. Θα μιλήσω για τη flexicurity, την ασφάλεια. Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον αυτό. Υπήρξε εισηγητής για το θέμα πριν από χρόνια και βρίσκω ότι ήταν τεράστια η πλειοψηφία που ψήφισε υπέρ του συστήματος αυτού. Έλα στα ασφάλεια, τρόπον την είναι αυτό. Συνεχίζει να το εξετάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο έχει πάψει να ενδιαφέρει. Ένας από τους λόγους είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλά κανείς για έλα στα ασφάλεια, εάν δεν υπάρχει ήδη ένα σύστημα πρώτης ασφάλειας. Δηλαδή, αν οι άνθρωποι είναι ασφαλεί τότε ε, είναι πολύ ελαστική. Αλλά το να είναι κανείς ασφαλής σημαίνει ότι του έχουμε εξασφαλίσει αξιοπρεπές εισόδημα και βασικά ε, εισοδήματα σε περίπτωση που είναι άνεργος, δηλαδή είναι επίδομα ανεργίας. Να μπορεί να, να ζητήσει επιπλέον εκπαίδευση, να μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά εργασίας. Να ξαναπώ ότι στη Δανία Έχουμε δύναμη εργατική 2,7 εκατομμύρια ανθρώπους περίπου, το 1 τρίτο. Αλλάζουν δουλειά κάθε χρόνο. Το 1 τρίτο. Οι άνθρωποι στη Δανία λένε δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά πια, θα κάνω μια άλλη. Δεν είναι πρόβλημα, διότι έχουν επίδομα ανεργία και μπορούν να ζήσουν από αυτό για ένα-δυο μήνες. Και μετά βρίσκουν άλλη δουλειά. Ξέρω όμως ότι αυτό δεν είναι το σύστημα σε πολλές από τις άλλες χώρες. Έχουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι. Και λέμε μετά ότι ο κόσμος στην αγορά εργασίας πρέπει να είναι πιο ε, ελαστικός. Με 20 εκατομμύρια ανέργους πώς να είναι πιο ελαστική. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα σύστημα κοινωνικής πρόνοιας ώστε να φροντίζουν τους ε, ευάλωτους. Αυτό που αναφέρατε κι εσείς. Αυτό είναι απαραίτητο. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα επιληθεί με αυτές τις πρακτικές. Πρακτικές ε, που ε, θα αναλυφθούν σε επίπεδο εταιρεία. Η κοινωνική εταιρεία είναι αυτή που πρέπει να βρουν λύση στα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο και πραγματικά είμαι υπέρ μια τέτοια επιλογή. Αν θέλουμε όμω ο κόσμο να είναι ελαστικό, πρέπει να του δώσουμε πρώτα ένα σύστημα ασφάλεια. Τότε θα γίνουν πραγματικά ελαστικοί. Ευχαριστούμε πολύ όλοι. Ο λόγο στο κοινό για ερωτήσει, σχόλια. Απλώ θα σα παρακαλέσω να μα λέτε το όνομά σα και από ποιον οργανισμό ε, προέρχεστε. Ευχαριστώ. Μπέγκαν από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ στον Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλο αυτό το θέμα για τη βιώσιμη εργασία πραγματικά με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και θέλω να σχολιάσω το θέμα των γυναικών μάνατζερ, στη δίκηση δηλαδή, όπου βλέπουμε να επιτελείται πρόοδος, αλλά έχουμε και διάφορα κενά και ελλείψεις, ένα ολόκληρο κατάλογο και εκεί το Ίδρυμα καλό θα ήταν να σταθεί λίγο σε αυτό, το πώς προχωράει η διάσταση ευθυγράμμισης του φίλου. Ε, οι γυναίκες στο management λοιπόν. Ε, οι γυναίκες αυτές έχουν λιγότερες πιθανότητες να κάνουν παιδιά από ότι άντρες manager και κάποιος μάλλον στο σπίτι πρέπει δεν θα τις βοηθά στο σπίτι. Επίσης το χάσμα στις πληρωμές της αμοιβές μεγαλώνει, μεγαλώνει στο μέσο όρο σε πολλές χώρες. Όταν είναι κανείς ε, ακριβώ κάτω από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο, εργασιακέ συνθήκε σχετίζονται με όλο αυτό ε, και πολλέ φορέ είναι και τελείω ε, δύσκολε ε, και μάλιστα με το που περνά μια γυναίκα τη γυάλινη οροφή την κρυστάλλινη ροφή φτάνει στο κρυστάλλινο, στην κρυστάλλινη άβυσο μπροστά τη. Δηλαδή πρέπει να αντιμετωπίσει ευθύνε και φιλόδοξα προγράμματα που είναι ακόμη πιο δύσκολα. Οι γυναίκε, μάλιστα, μάνατζερ, πολλέ φορέ βρισκόνται σε δημόσιε υπηρεσίε και με τεράστια πίεση στην υγεία, την εκπαίδευση και τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Οι ικανέ γυναίκε λοιπόν προχωρούν στο management αλλά για να έχουν βιώσιμες διαδροδρομίες και βιώσιμη παροχή υπηρεσιών εμείς προς αυτές, πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά τις εργασιακές τους συνθήκες. Όχι απλώς να θεωρούμε ότι είναι μια προνομιακός ελίτ γυναικών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Άλλα σχόλια ή ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Εμιλοίζα Πρίστα από την Πορτογαλία. Και έχω μια ερώτηση προς την ε, Τατιάνα αναφέρατε την ανάγκη να αναγνωριστεί η αξία της απλήρωτης εργασίας και να είναι αυτό ε, πολιτικός στόχος τη άμεση δηλαδή εργασίας. Η ερώτησή μου είναι πώ σκέφτεστε να το πετύχετε. Μπορείτε να μα πείτε περισσότερα για την κατεύθυνση και τι εντάσει που μπορεί να δημιουργούνται στην πολιτική συζήτηση για την αναγνώριση τη δουλειά αυτή των φροντιστών Ευχαριστούμε. Εάν υπάρχει τρίτη ερώτηση ή σχόλιο, το δέχομαι. Μετά όμως όχι. Ναι. Ρόναλντ Γιάνσεν. Μας απασχολούν κάποια από τα αριθμητικά στοιχεία εδώ, γιατί είπα το 85% των εργαζομένων είναι ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, οπότε ε, εάν 85% είναι ικανοποιημένοι, και το είπαμε αυτό το πρωί, πώ το απόγευμα λέμε ότι 25% των εργαζομένων πιστεύουν ότι η δουλειά του δεν είναι καλή για την υγεία του. Οι αριθμοί δεν φαίνεται να συμφωνούν. Έχετε κάποιο σχόλιο. Ευχαριστούμε. Να δώσω το λόγο στην Τατιάνα. Θες να απαντήσεις. Να απαντήσω, να σχολιάσω μάλλον το, το, τη δήλωση της Βλαντιμίρα. Όχι άλλη ρύθμιση. μέρος των αριθμίσεων είναι οι που είναι πιο ευέλικτες στο στην προσπάθεια ρύθμισης του επαγγελματικού βίου. Είναι θέμα πολιτικής θέσης βεβαίως. Από την αριστερή πτέρυγα του Κοινοβουλίου εγώ, γνωστό είναι σε όλους και πρέπει να το πω ότι Είμαστε υπέρ των κοινωνικών υποθέσεων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Σίγουρα υπάρχει μια έλλειψη ισορροπίας στη ρύθμιση εμπορικών ζητημάτων, αλλά όχι ελάχιστον μισθών λόγου χάρη. Και άλλα σημαντικά ζητήματα, άλλες πτυχές που είναι σημαντικές για τον κοινωνικό βίο των ανθρώπων. Αυτό είναι ο λόγος που κάποιες φορές λαμβάνονται αποφάσεις και καταλήγουμε σε αποτελέσματα όπως το Brexit. Δεν μπορεί να είναι κανείς ημιαγκαίος. Ή θέλει νομοθεσία ή δεν θέλει. Και κάθε χώρα θα χαράξει τη δική της πορεία. Όπως ε, προείπα, αυτή είναι η θέση μας. Όλο και περισσότερο οι πολιτικές ομάδες της δεξιάς, τέργας και το Κοινοβουλίο συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει περισσότερη ρύθμιση σε κοινωνικά ζητήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, το σχολείο σα για την άμεση εργασία, έχουμε προτείνει πολλά. Δεν μπορώ να τα συνοψίσω. σω να διαβάζατε την έκθεσή μα. Υπάρχει μια σειρά από προτάσει την, με αφορμή την οδηγία των φροντιστών. Βεβαίω μπορεί να έρθει ω νομοθετική πρόταση από την Επιτροπή, θα το σκεφτούμε Και θα δούμε τι διαδικασία θα ακολουθήσουν στην επεξεργασία της πρότασης. Πάντως, οι υπηρεσίε φροντίδα θα πρέπει να επιλογίζονται λόγω χάρη στον τελικό απολογισμό μια σύνταξη. Είναι μια πρώτη ιδέα. Κάπως έτσι θα να χωρίσουμε σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Τατιάνα, έχεις ένα λεπτό για να απαντήσει. Στα αυτού του είδου τη μελέτη για τι ε, εργασιακέ συνθήκε, η ικανοποίηση είναι ένα κριτήριο. Αλλά πάντοτε βρίσκει κανεί ψηλά ποσοστά ε, ικανοποίηση. Είναι μια ερώτηση και ο κόσμο την να απαντάει θετικά. Εάν όμω κανεί αρχίσει και το σκαλίζει, εκεί είναι που βρίσκει ζητήματα ε, επιμέρου που μπορεί να προκύπτουν και δεν είναι αντιφατικό λοιπόν αυτό που εντοπίσατε. Προσπαθούμε να δούμε τα αριθμητικά στοιχεία, χωρίς να μένουμε στην ικανοποίηση, αλλά προχωρούμε και βαθύτερα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς ο κόσμος αισθάνεται για τις εργασιακές του συνθήκες. Και μετά ενώνουμε τα κομμάτια του παζλ. Και Κολέτ, να προσθέσω κάτι και να πω ότι να ξέρεις θα κάνουμε μια ειδική ανάλυση για τις γυναίκες μάνατζερ και ήδη έχουμε ξεκινήσει. Θα έχουμε και περισσότερα αποτελέσματα σύντομα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις σημαντικές πληροφορίες που περιλαμβάνει το έγγραφο αυτό. Νομίζω η συζήτηση σήμερα ήταν πλούσια, έθεσε πολλά σοβαρά ζητήματα και νομίζω ότι θα μπορέσει να ενσωματωθεί πολύ καλά στην πολιτική μας συζήτηση για τις σχετικές αποφάσεις. Είναι τέσσερις, ευτυχώς ε, προλάβαμε στην ώρα μας. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και το κοινό μας. Καλησπέρα σας. Θα προσπαθήσω κι εγώ να μιμηθώ την προκάτοχό μου και τις καλές επιδόσεις ό,τι αφορά την τήρηση του χρόνου. Γι' αυτό παρακαλώ καθίστε για να συνεχίσουμε και σας ευχαριστώ για το κουράγιο σας γιατί πραγματικά μείνατε μέχρι το τέλος ε, τη ε, του τελευταίου πάνελ. Φανταζόμουν, φοβόμουν ότι είμαστε περισσότεροι στο πάνελ από ό,τι στην Ομίγυρη. Είμαι ο Χέρμαν Φόγκ, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Eurofound και εργάζομαι για τα βελγικά συνδικάτα. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, γιατί άκουσα τα αποτελέσματα της νέας επισκόπησης για τις εργασιακές συνθήκες και βλέπουμε ότι έχουμε ένα νέο ορόσημο σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των εργασιακών συνθήκων και την ε, άντληση πολύ χρήσιμων στοιχείων για τους κοινωνικούς εταίρους, πολιτικούς. Ήδη η έρευνα αυτή δίνει λαβή και τροφή για πολλή συζήτηση γιατί πολύ συχνά υπάρχει διάσταση σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα. Εγώ χαίρομαι ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Eurofound και μέλος και της ε, Συμβουλευτικής Επιτροπής. Είμαι προνομιακός παρατηρητής πολλές φορές και χαίρομαι πώς αναπτύσσεται αυτή η επισκόπηση. Θα ήθελα τώρα στο πάνελ αυτό να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο στον τρόπο χρήσης ε, των στοιχείων της επισκόπησης στην πολιτική συζήτηση πώς θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία για την ποιότητα της ζωής, πώς χρησιμοποιούνται και τι δυνατότητα υπάρχει για μια νέα ατζέντα για την ποιότητα της εργασίας, για την εργασιακή ζωή και πώς εφαρμόζονται οι διάφορες προσεγγίσεις ε, για τα θέματα αυτά. Θα παρουσιάσω τα μέλη του πάνελ ε, και θα μας πούν ε, πώς καθημερινά χρησιμοποιούν ε, τα απορίσματα του Eurofound. Θα ξεκινήσουμε με την Barbara Gerstenberger, που είναι συντονιστή στη διεύθυνση της Eurofound και θα μας πει πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα της επισκόπησης αυτής του Eurofound από τους πολιτικούς ηθήνοντες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Χέρμαν. Μου έκανε τις πρώτες συστάσεις. Ε, λέγομαι Μπάρμπαρα Γκέρστεμπεργκερ και είμαι συντονίστρια στο διευθυντήριο της Eurofound. Οπότε είμαι εξοικειωμένη όχι μόνο με την επισκόπηση για τις εργασιακές συνθήκες στην Ευρώπη, αλλά και με άλλες έρευνες και μελέτες της Eurofound είμαι εξοικειωμένη. Έχω μια γενική επισκόπηση όλων αυτών των μελετών και ερευνών. Τώρα τι γνωρίζουμε, όπως ρώτησες, για τη χρήση των αποτελεσμάτων της επισκόπησης αυτής για τις εργασιακές συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς χρησιμοποιούνται, πώς αξιοποιούνται. Από του ε, πανελίστε που ακούσαμε μέχρι τώρα, από εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ευρωβουλευτέ, συχνά ακούσαμε και χαιρόμαστε γι' αυτό πόσο πολύ χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα, τα πορίσματα των μελετών μα. Και ένα από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στη συζήτηση για, για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν τα πορίσματα του Eurofound. Μάλιστα και ζητήθηκε από τη Eurofound να επενδύσει ακόμη περισσότερο στην παρακολούθηση τέτοιων εργασιακών συνθήκων στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρθηκε η έκθεση για την εξασφάλιση εργασιακών συνθήκων που να προωθούν το συνδυασμό εργασίας και προσωπικής ζωής. Εκεί Επίσης απευθυνθήκε έκκληση στο Eurofound να συνεχίσει ε, την παρακολούθηση και τη διερεύνηση των εργασιακών συνθήκων στην Ευρώπη. Είναι δύο πρόσφατα παράδειγμα που δείχνουν πόσο συστηματικά χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματα των μελετών μας, της επισκόπησής μας σε έγγραφα πολιτικής. Και μάλιστα το 2010 στην πέμπτη έκθεση, μέχρι τα τέλη του 2013 γνωρίζαμε ότι πάνω από 50 έγγραφα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιούσαν τα δικά μας στοιχεία, τα στοιχεία του Eurofound για την, ε, τις κοινωνικές εξελίξεις ε, και στην Ευρώπη. Αλλά αναφέρθηκε ε, και η χρήση των στοιχείων αυτών από, το ΟΣΑ, από τον ΩΣΑ από τη ΔΟΕ και άλλοι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούν τα στοιχεία μας. Αλλά και το Ινστιτούτο των, δύο φίλων στο Βίλνιους χρησιμοποιεί επίσης τα στοιχεία της δικής μας επισκόπησης μας για να συμπληρώσει τον δικό τους δίκτυο ισότητας των φίλων. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Αυτά σας αρκούν για το πώς αξιοποιείτε τα συμπεράσματά μας. Μάλιστα. Περνάμε τώρα στον κύριο Τον Μπέβερ, στον παρακαθήμενο, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, ΕΜΚΟ. Θα μας ε, παρουσιάσει στην συντομία την Επιτροπή του και θα μας πει πώς σχετίζεται το έργο της Επιτροπής του με τα πορίσματα της επισκόπησης του Eurofound. Όπως ξέρετε, η ΕΜΚΟ είναι το κύριο συμβουλευτικό σώμα για θέματα απασχόλησης ε, του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και ε, κυρίως ως προς το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Παρεβαίνουμε σε σημαντικά ορόσημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδιαίτερα κατά τη σύνταξη των ειδικών συστάσεων αναχώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκεί ε, παρέχουμε συμβουλέ προκειμένου να τροποποιηθούν ε, οι στάσει αυτέ πριν τι υιοθετήσει του Συμβούλου. Και μάλιστα χθε ε, είχαμε την κοινή έκθεση για την Ευρωζώνη, το σχέδιο συστάσεων και όλα αυτά τα έγγραφα τα εξετάσουμε στο, την επόμενη Δευτέρα, ώστε στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων να, να αξιοποιηθούν για να αποκρισταλωθεί θέση του Συμβουλίου. Έχω μια πολυμερή ε, προσπάθεια επισκόπησης ε, και έρευνας και τη συμπληρώνουμε με ένα αναλυτικό έργο σε μια τεκμηριωμένη προσέγγιση ε, για την διαμόρφωση της θέσης της πολιτικής απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και εκεί χρησιμοποιούμε το, τα πορίσματα της Eurofound και μάλιστα η ιδιαίτερη επισκόπηση των ρωσιακών συνθηκών είναι πολύ χρήσιμη στο δικό μας έργο γιατί η έρευνα αυτή, η επισκόπηση αυτή παρέχει πληροφορίες για το κοινό αναλυτικό ε, πλαίσιο και το πλαίσιο των επιδόσεων. Ε, και έτσι λαμβάνουμε υπόψη το θέμα της ποιότητας εργασίας και πώς επηρεάζει την ε, εργασία γενικώ. Τώρα στο μέλλον. Θα έχουμε φυσικά και συμμετοχή στη συζήτηση για τον κοινωνικό πυλώνα. Ήδη έγιναν πολλέ αναφορέ σήμερα για το θέμα του κοινωνικού πυλώνα και εκεί θα χρειαστούμε ε, τεκμηριωμένη συζήτηση, εμπεριστατωμένη και γι' αυτό θα πρέπει να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία της επισκόπησης του Eurofound. Εμείς, η Επιτροπή Απασχόλησης, ε, σε μια κοινή γνωμοδότηση με την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, δεν ε, ε, έχουμε υποβάλει στο Συμβούλιο και μάλιστα έχει εγκριθεί. Θεωρούμε ότι ο κοινωνικός πυλώνας θα πρέπει να δράζεται στο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Και μάλιστα έχει αποδείξει την ευελιξία του αυτός ο μηχανισμός και μάλιστα καταλήγει σε απτές αλλαγές πολιτικής ε, και πιο προσάρμοστε στις αλλαγές τη απασχόλησης. Φυσικά, νέα αντιμετώπιση δεν χωρεί εδώ, λόγω των ιδιαιτεροτήτων. Και ένα τμήμα των αρμοδιοτήτων είναι κοινοτικό. Γι' αυτό και ο κοινωνικός πυλώνας θα πρέπει να βελτιώσει και να ενισχύει τους μηχανισμούς και τα εργαλεία που έχουμε και έτσι θα διαμορφώσουμε και ένα μελλοντικό πρόγραμμα εργασιών κοινωνικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το έργο αυτό λαμβάνουμε υπόψη και τις εργασίες στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας και στον ΩΣΑ, ώστε να επιτύχουμε την σύγκληση προς τα πάνω που θέλουμε. Με σεβασμό φυσικά των εθνικών αρμοδιοτήτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γι' αυτό, κύριος Στέφανος Καρπέτα τώρα, θα σας θέσω την ίδια ερώτηση. Μπορείτε σύντομα να πείτε τι κάνετε στον ΩΣΑ και πώ αξιοποιείτε τι μελέτε του Eurofund στη δουλειά σα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σα, κύριε και κύριοι. Το όνομά μου πράγματι είναι Στέφανο Καρπέτα και εργάζομαι για την απασχόληση, την εργασία και τι κοινωνικέ υποθέσει των ΩΣΑ με την ε, ε, εφαρμογή των ε, εργασιακών πολιτικών, την μετανάστευση και την υγεία και τέτοια θέματα. Είναι χαρά μου που είμαι σήμερα εδώ στη διάσκεψη αυτή για να συζητήσουμε τα βασικά θέματα της έκτης έρευνας για την ε, απασχόληση. Νομίζω ήταν ενδιαφέροντα όσο υπόθηκαν στις προηγούμενες φάσεις ε, της, διάσκεψης, της σημερινής μας συνεδρίασης. Να σας πω τι κάνουμε εμείς στη δουλειά μας στον ΩΣΑ. Έχουμε αναπτύξει ένα πλαίσιο για την ποιότητα της εργασίας που χρησιμοποιεί διεξοδικά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα της μελέτης για τις ευρωπαϊκές εργασιακές συνθήκες. Η ποιότητα της εργασίας ε, αναφέρθηκε στην ε, στρατηγική για την εργασία του ΩΣΑ, το βασικό στρατηγικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να, για να αξιολογήσουμε τις πολιτικές και τις αγορές εργασίας των κρατών μελών. Ε, θα ξεκινήσουμε σύντομα τη μελέτη για το 2018. Κοιτάζουμε λοιπόν για καλύτερε δουλειέ, αλλά πλευρά αυτή δεν είχε προχωρήσει πολύ. Το πλαίσιο για την οδηγία των ε, ε, αγορών εργασίας κοιτάει τις επιδόσεις όλων των μελών του ΩΣΑ, όχι μόνο πώς χάνονται ή δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά και την ποιότητά τους. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί στη συστηματική μας αξιολόγηση των ε, πολιτικών για τις αγορές εργασίας, αλλά και με σκοπό να εντοπιστούν πολιτικοί στόχοι για να έχουμε συγκεκριμένη ποσότητα αλλά και ποιότητα θέσεων εργασία στην Ευρώπη. Στην επισκόπηση για την απασχόληση δημοσιεύσαμε ήδη δύο κεφάλαια, αλλά ήρθαν και οι Υπουργοί Εργασία στον ΩΣΑ, οι οποίοι σε μια σύντομη διασκεψή του ε, έδωσαν εντολή στον ΩΣΑ να αναπτύξει το σχετικό στρατηγικό του πλαίσιο. Είναι πολύ διάστατο το πλαίσιο αυτό. Κοιτάζουμε την ποσότητα, την ποιότητα, την συμμετοχικότητα τη αγορά εργασία και την ανθεκτικότητά τη. Αυτή είναι η δική μα η ατζέντα. Και γι' αυτό η δουλειά του Eurofund για την ποιότητα τη αγορά εργασία ειδικά πραγματικά τροφοδοτεί την δική μα. Ευχαριστούμε και τώρα η Μανουέλα Τομέη. Επίση, η διερώτηση και σε εσά. Θα μπορούσατε να συστηθείτε για να μας πείτε πώς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας αξιοποιείται τη δουλειά του Eurofund. Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση από Eurofund. Είμαι η Μανουέλα Τομέη, Διευθύντρια για τις Συνθήκες Εργασίας και την Υπηρεσία Ισότητας, το οποίο είναι γνωστό με το ακρόνιμο Work Quality, όπως καταλαβαίνετε από τον τίτλο μας, η βελτίωση των συνδικών εργασία και άλλε πτυχέ στην ποιότητα τη εργασία είναι πραγματικά στο επίκεντρο των όσων κάνουμε. Είναι μια κύρια διάσταση τη εξωπρεπού εργασία στον ε, Παγκόσμιο Οργανισμό, όπου κοιτάζουμε και την ποσότητα και την ποιότητα των θέσεων εργασία. Πραγματικά Έτσι όπως ε, ε, καταβάλουμε προσπάθειες στον ΩΣΑ, ο στόχος είναι να εντοπίσουμε όχι μόνο τάσεις, αλλά και τι θα μπορούσε να οδηγήσει τους ε, υπεύθυνους φορείς να έχουν τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στις εργασίες, χωρίς να θέσουν κινδύνο την ασφάλεια Τη αγορά εργασία. Κοιτάζουμε δηλαδή να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ τη ποιοτητα και τη ασφαλεία. Έχουμε καταλήξει σε μια σειρά από δραστηριότητε λόγω αυτού, του προβληματισμού. Θα δώσω απλώ ένα παράδειγμα. μόλι δημοσιεύτηκε και άλλη μία θα δημοσιευτεί σύντομα μια μελέτη για το πώ οι αλλαγέ στη διοργάνωση της παραγωγής και του εργατικού δυναμικού στον κόσμο επηρεάζει τις εργασιακές συνθήκες. για την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Οι ποιοτικέ θέσει εργασία μα απασχολούν από τη σκοπιά τη πρόνοια και τη κάλυψη των εργαζομένων, αλλά και τι επιπτώσει υπάρχουν για τι επιδόσει των επιχειρήσεων. Πολύ σύντομα, Θα έχουμε και τη δημοσίευση της έκθεσης για τους ε, μισθούς παγκοσμίω με τάσεις ε, που μελετώνται με βάση κάποιους συγκεκριμένου ε, συντελεστές υπολογισμού των μισθών. Το μέσο όρο, την κατανομή τους, σε όλους τους εργαζομένους. Και επίσης θα δούμε τις εξελίξεις της μισθολογικής πολιτικής, την εκπαίδευση και την ισότητα. συνειδητοποιούμε ότι η εξέταση των μισθών και των απολαβών είναι μια σημαντική διάσταση της έννοιας της ποιότητας στην εργασία. Σίγουρα δεν είναι αρκετή. Λόγω της ευρύτητας των πολλών άλλων θεμάτων που άπτονται του θέματος αυτού, γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το Eurofund με σκοπό από κοινού να προσπαθήσουμε να επεκτείνουμε το γεωγραφικό πεδίο των μελετών μας, της ε, μελέτης εργασιακών συνθήκων του Eurofund. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δραστηριοποιούμαστε σε τρεις επιπλέον χώρες, την Κίνα, τις Ηνωμένε Πολιτείες, Αμερικής και την Κορέα. Ρωτήσατε πώς χρησιμοποιούμε τη μελέτη αυτή. Σε καθημερινό επίπεδο τη χρησιμοποιούμε. Και θα ήθελα να δώσω και ένα παράδειγμα. Συγκριτική δουλειά που αυτή τη στιγμή διεξάγουμε ως μέρος των, της των διεθνών προτύπων για την παρενόχληση ε, και την, ε, τον εκφοβισμό στον χώρο εργασίας. Άρα, να στραφώ ξανά στην Μαρίτα. Μίλησες και το πρωί. Μπορεί να μας περιγράψει λίγο. Εσεί στη δουλειά σα πώ χρησιμοποιείτε την έρευνα αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, πάλι, πάλι εδώ είμαι. Για όσους ήρθαν τώρα, είμαι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας απασχολεί λοιπόν, ε, απασχολούν τα θέματα απασχόλησης και τα κοινωνικά και για να απλοποιήσω τα πράγματα. Το Eurofund θα έλεγα είναι ε, δικό μας. Γιατί η Επιτροπή ε, Απασχόλησης έχει... Εντάξει, υπάρχουν διάφοροι φορείς που σχετίζονται μεταξύ μαζί μα. άμεσα και το Eurofund θα έλεγα πω είναι το ερευνητικό μας Ινστιτούτο. Αυτό σημαίνει ότι Ε, δύσκολα μπορούμε να είμαστε κατά πραγμάτων που ε, διαπιστώσαμε ότι έπρεπε να μας απασχολούν. Δεν είχαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που παράγει το Eurofund. Ε, δεν θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε για αυτά τα οποία θέλουμε να πετύχουμε. Τυχαίνει καμιά φορά να ζητάμε από το Eurofund νούμερα και στοιχεία αλλά θα έλεγα ότι συνήθως οι περισσότερες από τις εκθέσεις είναι το αποτέλεσμα ερευνών των ερευνητών του Eurofund που ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς ε, το θεσμικό μας όργανο θέλει να μάθει περισσότερα και βεβαίω θα έχουμε κάποια αποτελέσματα στο πολιτικό επίπεδο, αλλά δεν λέμε ότι πρέπει να κάνεις αυτό. Όχι, όχι. Είναι μια πάρα πολύ στενή ε, σχέση και με την Επιτροπή μας και με τους άλλους επιστημονικούς φορείς, αλλά Θα έλεγα λοιπόν ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία και εκθέσεις της Eurofound. Αυτή είναι η έκθεση που παρουσίασε η Eurofound. Αυτή είναι η έκθεση ακριβώς που έδειξε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτά τα οποία συζητάμε δηλαδή από το πρωί και συζητάμε ακόμα τον αντίκτυπο του κοινωνικού διαλόγου και συχνά τα συγκεκριμένα αποτελέσματά του, που είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Και ήταν ευκολότερο έτσι να περάσουν την κρίση και χωρίς να καταλήξουν σε μια απελπιστική κατάσταση. Γνωρίζουμε πως ε, πολλά κράτη-μέλη δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο, αλλά μπορούσαν και είμαστε οπωσδήποτε σε πολύ καλύτερη μοίρα από αυτούς που δεν είχαν ποτέ ακριβώς ε, τους κοινωνικούς εταίρους και τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για εμάς στις συζητήσεις με άλλες επιτροπές στην Οικονομική Επιτροπή όταν συζητάμε επενδύσεις, όταν συζητάμε το πώς θα βγούμε από αυτή την κρίση και θα έχουμε ισχυρά κράτη-μέλη. Και αυτή η έκθεση είναι ακριβώς παράδειγμα του πώς χρησιμοποιούμε το Ίδρυμα αυτό πώς συζητάμε δηλαδή και το πώς ε, βρίσκουμε μια ατζέντα η οποία ακριβώ μετά από λίγο αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να ακολουθεί. Έτσι γίνεται λοιπόν με την έρευνα και την πολιτική με σεβασμό ένας τον άλλον. Και ταυτόχρονα ε, μια επικοινωνία θα έλεγα η οποία να μας εμπνέει και τελικά καταλήγει σε χρήσιμα συμπεράσματα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα δεύτερο γύρο και μετά έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις. Να επανέλθω στην Μπάρμπαρα, ίσως, να σας ρωτήσω. Ε, μια ίσως ενοχλητική ερώτηση. Αν δείτε την έρευνα Ποια είναι τα βασικά διδάγματα πολιτικής ε, κατά την άποψή σας. Είδαμε ότι ήδη κάποιοι συνάδελφοι ε, μίλησαν για την ισορροπία ε, προσωπικής και κοινωνικής ζωής. 81% είναι ικανοποιημένοι, το 19% είναι ήδη αρκετά εκατομμύρια που δεν είναι ικανοποιημένοι. Εσείς ως αντικειμενικοί τι άποψη έχετε Ευχαριστώ. Πριν απαντήσω. Να πω βέβαια στη Μαρίτα πως είναι πάρα πολύ ευχάριστα αυτά τα οποία λέτε, ότι το Eurofound είναι δικό μας. Θέλουμε να είμαστε το ερευνητικό σας κέντρο και να σας δίνουμε τα στοιχεία που θέλετε ε, και για την χάραξη πολιτικής στο μέλλον. Ε, διαμαρτύρομαι εγώ και εκ μέρους των ε, τριμερών διαπραγματεύσεων είναι και δικό μας. Λοιπόν, ναι, ναι, ακριβώς. Ε, είμαστε το ερευνητικό Ίδρυμα των Κοινωνικών Εταίρων. Και στηρίζουμε βεβαίως και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα σας για τα μηνύματα της πολιτικής Νομίζω πω ε, είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο και δεν θέλω να επανέλθω σε κάτι που ανέφερε νωρίς. νωρί. Είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε. Είναι πραγματικά κάτι που θα θέλαμε να το κρατήσετε ως συμπέρασμα το ότι καμία δουλειά δεν είναι τέλεια και ότι οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να βελτιωθεί σε κάποια από τις 7 ε, διαστάσεις που αναφέραμε. Και βεβαίως ελπίζω να μην βαρεθήκατε, μιλήσαμε για τα προφίλ αυτά ποιότητας εργασίας, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο ίσως να γίνουν κατανοητά, οπότε ε, εντάξει επαναλαμβάνομαι αλλά να τα ξαναπώ. Να ακούσουμε τις πολύ έτσι, απαιτητικές δουλειές που ε, εκ πρώτης μοιάζουν πολύ καλές, πολύ ευχάριστες, το, το μπλε χρώμα αν θυμάστε. Αλλά από τους 7 δείκτες υπάρχουν δύο δείκτες που δεν τα πάνε καλά. Το ένα είναι η ένταση εργασίας, γιατί έχουν υψηλό μεγάλες απαιτήσεις, ε, μεγάλες ταχύτητες και βεβαίως ποιότητα. Ε, πολλές ώρες, ε, πολλή δουλειά εκτός του κανονικού ωραρίου, οπότε ακόμα και αν τις λέμε δουλειές έτσι υψηλών απαιτήσεων και απολαβών, έχουν προβλήματα. Επίσης, οι δουλειές, οι στρωτές ας πούμε, και πολλές ε, πάλι εκεί πέρα δυνατότητες στους 5 από τους 7 δείκτες, αλλά και εκεί πέρα δεν υπάρχει διακριτική ευχέρεια και ε, χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων και ε, βεβαίως απολαβών. Οπότε και πάλι καλές, αλλά με κάποιους, κάποιες βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν. Οπότε, αν να δώσουμε κάποια προτεραιότητα βεβαίως, εγώ θα έλεγα, κοιτάξτε το προφίλ που έχουμε βρει εκεί, γιατί ε, εκείνο δεν έχει καθόλου μπλε κομμάτια, τετραγωνάκια, είναι όλο πορτοκαλί, οπότε απαιτούνται βελτιώσει σε όλους αυτούς τους τομείς. Ή αλλιώς πρέπει να σκεφτούμε πολιτικές ε, στην που επιτρέπουν στον κόσμο να φύγει από αυτές τις δουλειές χαμηλής ε, ποιότητας. Και βεβαίω ε, αυτό μπορεί να είναι θετικό ή αρνητικό, στο προφίλ αυτό βρίσκουμε πολύ κόσμο με προσωρινά συμβόλαια. Αυτό σημαίνει ότι είναι βεβαίως μπορεί να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για πιο ποιοτικέ δουλειέ. Αλλά αυτό οπωσδήποτε δεν θα γίνει αυτομάτως. Και βεβαίω πάλι θα απαιτηθεί κάποια δράση από την πλευρά τη πολιτική. Το καλό είναι αν δείτε την ποιότητα των θέσεων εργασία και διακρίνουμε τις 7 διαστάσεις με τους 7 δείκτες, Έχουμε πολλές αφετηρίες αν θέλουμε να βελτιώσουμε κάτι. Βεβαίω αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιο μαγικό ραβδάκι, αλλά και βέβαια υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που αφορούν το χρόνο εργασίας, την ε, ισορροπία με την προσωπική ζωή. Αυτό νομίζω σε γενικές γραμμές είναι θετικά ναι. Just ε, return to you, Marita, back again. Marita, ε. ξαναστρέφομαι προς εσένα γιατί η Μπάρμπαρα μας εξήγησε τι γίνεται με τις εργασίες χαμηλής ποιότητας και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι συγκρίθηκαν με τους ψηφοφόρους του Τραμπ, αυτούς που ψήφισαν υπέρ του Brexit. Θεωρείς ότι οι υφιστάμενες ευρωπαϊκές πολιτικές είναι στο ύψος των προσδοκιών αυτών των ε, χαμηλόμισθων ε, εργαζομένων ή αυτών που απασχολούνται σε εργασίες κακής ποιότητας, χαμηλής ποιότητας. Η Μαρίτα. Φυσικά θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά και να βελτιώσουμε τις προσπάθειές μας και τα αποτελέσματα. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε την ε, συνδιάσκεψη κάπως πεσμένη ψυχικά, κάπως ε, απογοητευμένη και διαπιστώσαμε ότι πολλοί άνθρωποι είναι οργισμένοι, αγανακτισμένοι και έχουν και σωστά πολλές φορές την αίσθηση ότι κανείς δεν νοιάζεται για τη, για ποιότητα ζωής τους ε, ή για την ποιότητα της, του εργασιακού τους περιβάλλοντος και δημιουργήθηκαν συστήματα ή συνθήκες που ενισχύουν την αντιπαράθεση μεταξύ των ανθρώπων ε, αντί να δημιουργούνται προϋποθέσεις για συνεργασία για την καταπολέμηση των κοινών προβλημάτων. Επίσης αναφέρθηκε το κοινωνικό ντάμπινγκ και την ανάγκη μιας ε, λειτουργικής οδηγίας για τους αποσπασμένους εργαζομένους, ώστε να μην έχουμε ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εργαζομένων και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια κούρσα προς τα κάτω για χαμηλότερους μισθούς ή ε, χειρότερη ποιότητα σε επικίνδυνα εργασιακά περιβάλλοντα. Θα πρέπει ο ανταγωνισμός να μην γίνεται μεταξύ μας, αλλά με άλλους εταίρους του κόσμου. Ε, και να είμαστε πραγματικά καλοί σε αυτό που κάνουμε. Αλλά θα τα καταφέρουμε αν ε, λοφαγωνόμαστε και αν ε, η αντιπαράθεση είναι εσωτερική, μεταξύ του Βορρά και του Νότου για παράδειγμα, της Ανατολής και της Δύσης. Θα πρέπει να υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μας, όχι αντιπαράθεση. Επίσης, ε, θα θυμάστε ότι ο κύριος Πυρίσκη, από την ίδια πολιτική ομάδα με μένα, μίλησε για την παραγωγή που έχουμε πολύ μορφωμένων ανθρώπων από την Ανατολική Ευρώπη που εξάγονται προς τις άλλες χώρες Ευρώπης όπου έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο και καλύτερες αμοιβέ. Ενώ ταυτόχρονα έχουμε εξαγωγή και άλλων ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να δεχτούν οποιαδήποτε δουλειά, όσο χαμηλοαμοιβόμενοι και αν είναι, μόνο και μόνο για να βρουν μια θέση απασχόληση. Είναι τόσο απελπισμένοι. Και υπάρχει αυτή η κίνηση μονόδρομη από την Ανατολική Ευρώπη προς τη Δυτική. Αν δεν βρούμε τρόπο να εξορροπήσουμε τα πράγματα, τέτοιου είδους συγκρούσεις θα μας οδηγήσουν σε μια κατάσταση ε, Donald Trump σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κανείς δεν είναι στο απειρόβλητο της μυσαλλοδοξίας ή επικίνδυνων συγκρούσεων μεταξύ των ανθρώπων. Θα πρέπει όμως να δούμε τι νόημα έχουν τα στοιχεία και να διευκολύνουμε αυτούς που έχουν υψηλή μόρφωση να παραμείνουν στις πατρίδες τους και να αξιοποιήσουν εκεί το δυναμικό τους και να μην πυροδοτούμε ρατσισμό, ρατσιστικά πάθη και αντιδημοκρατικά αισθήματα σε άλλες περιοχές Ευρώπης, βάζοντας τους εργαζόμενους σε μια κατάσταση όπου οι εργαζόμενοι της Δύσης βλέπουν περιφρονητικά ε, τους ε, εργαζόμενους της Ανατολικής Ευρώπης και θεωρούν ότι έρχονται και κάνοντας ντάμπιγκ των μισθών τους τρών τις θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια πλειοψηφία πρώτα εντό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά στο Συμβούλιο και να πούμε εντάξει, να έχουμε μια οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η υψηλά εξειδικευμένοι και πολύ μορφωμένοι ε, υπήκοοι της Ανατολικής Ευρώπης ε, να παραμένουν στις πατρίδες τους, γιατί οι χώρες ε, χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των υπηκών τους και μετά αυτοί σηκώνονται και φεύγουν και αναζητούν καλύτερο μέλλον σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Να μην νιώσουν οι συμπολίτε μας ότι είναι καταλημμένοι στη μοίρα τους, ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται. Πρέπει να βρούμε στοιχεία που να πείσουμε τους πολίτες ότι η Ευρώπη έχει νόημα. Αλλιώς θα έχουμε ε, πολύ απογοητευτικά αποτελέσματα, να μην πω ε, τρομερά αποτελέσματα ε, όπως αυτά των Αμερικανικών εκλογών. Γιατί τέτοιου είδους ε, φρικτά αποτελέσματα θα μπορούσαμε να έχουμε και εδώ για να μην πω και χειρότερα. Επίσης, στην Επιτροπή Απασχόλησης, πρωταρχή μας προτεραιότητα είναι η οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. ή η κατάσταση όπου σε κάποιες χώρες Ανατολικής Ευρώπης δεν ασκούνται οι ίδιες πιέσεις στις ε, επιχειρήσεις για την τήρηση κάποιων ε, περιβαλλοντικών κριτηρίων στον στο χώρο εργασίας. ακριβώς επειδή το οικονομικό πλαίσιο δεν είναι πολύ ευνοϊκό όπως στις υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και αν δεν την βρούμε θα έχουμε όλο και πιο πολλές ανειδίκευτες θέσεις εργασίας και όλο και περισσότερους αγανακτισμένους και εξοργισμένους συμπολίτε. Και αγανακτισμένοι θα είναι αυτοί που μένουν στην περιφέρεια της αγοράς εργασίας και που δεν μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας ή θα είναι εξοργισμένοι και αυτοί που είναι στην αγορά εργασία, αλλά υπό πολύ δυσμενεί συνθήκε. Ευχαριστώ για τα σχόλια. Πριν περάσουμε στη συζήτηση, να ρωτήσω τον παρακαθήμενο και πάλι. Τι κάνετε στην ΕΜΚΟ. Έχετε ένα σύστημα για την καταμέτρηση της εργασιακής ποιότητας. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε. Τα πορίσματά σας συνάδουν με αυτά της Eurofound, είναι αντιφατικά. Πώς λειτουργούν τα πράγματα και σε εσά στην ΕΜΚΟ. Όντως στην Επιτροπή Απασχόληση έχουμε μακρά παράδοση στο τομέα της ποιότητας στην εργασία. Εγώ το 2001 ξεκίνησα όταν πρότεινε κάτι τέτοιο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τότε η Επιτροπή Απασχόληση έδειξε μια σειρά δικτών για τις επιμέρους διαστάσεις που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που εγκρίθηκε τελικά από το Συμβούλιο. Και μάλιστα ήταν ε, ρηξικέλευθη αυτή η πρωτοβουλία τότε. Ήμασταν ίσως πρώτη διεθνής επιτροπή που είχε ένα τέτοιο κατάλογο. Στο μεταξύ βέβαια πολλά έχουν αλλάξει και πολλά άλλα θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανώσεις ε, έχουν δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα και αυτό μας χαροποιεί. Το 2013-2014 ενημερώσαμε τον κατάλογο με τους δείκτες μας και αποφεληθήκαμε από τις πληροφορίες της πέμπτης επισκόπησης του Eurofound για τις εργασιακές συνθήκες στην Ευρώπη και επίσης αξιοποιήσαμε και το έργο του ΟΣΑ. Σήμερα λοιπόν οι δείκτες μας που περισσότεροι στηρίζονται σε αυτή την επισκόπηση του Eurofound συμπεριλαμβάνονται πια στο αναλυτικό έργο μας ώστε ε, και το ευρωπαϊκό εξάμεινο να είναι μια τεκμηριωμένη διαδικασία και μάλιστα παρακολουθούμε και την, ε, τις επιδόσεις στην απασχόληση και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών ε, Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόληση τον περασμένο μένα και από τα στοιχεία της έκτης έκθεσης του Eurofound θα ενημερώσουμε και θα επικαιροποιήσουμε και τα δικά μας στοιχεία και τα, θα δούμε τι συμπεράσματα για τις περαιτέρω πολιτικές μπορούμε να αντιλήσουμε από την τελευταία αυτή έρευνα του Eurofound. Πάντως η επισκόπηση, όπως τη βλέπω τώρα, χρήζει μιας περαιτέρω ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων, κάτι που θα εμβαθύνει τις γνώσεις μας για το θέμα. Πάντως αυτό που βλέπω και που επιβεβαιώνει τα δικά μας συμπεράσματα πολιτικής, τα πιο πρόσφατα, Καταρχήν το σίγουρο είναι αυτό που είπαμε και στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα. Θεωρούμε ότι οι προτάσει ευρωπαϊκή Επιτροπής δεν λαμβάνονται όντως υπόψη τη διάσταση του φύλου. Και τα πορίσματα της επισκόπηση του Eurofound στοιχειοθετούν αυτή μας την επιφύλαξη και την ανησυχία. Δεν έχουμε ισότιμη αγορά εργασία και για τα δύο φύλλα στην Ευρώπη. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη το στόχο μα. Επίσης, ε, διαφορετικά είδη ε, θέσεων εργασίας, διαφορετικά είδη συμβάσεων και ρευστότητα που υπάρχει. Ακόμη και ερωτηθέντες στην επισκόπηση, πολλές φορές ε, έχουν δυσκολίες στο να αυτοπροσδιοριστούν ως αυτοπασχολούμενοι, ως μισθωτοί. Ε, είναι περίπλοκοι μερικές φορές οι συμβασιακοί όροι. Και Γι' αυτό και λέμε ότι ο κοινωνικός πυρολόνας θα πρέπει να είναι οραματικός, να μην προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα του παρελθόντος, αλλά να ατενίσει το μέλλον και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Πολλές τις αναφέραμε και σήμερα. Και είναι πολύ πιο πολύμορφες πια οι εργασιακές σχέσεις. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Κάτι άλλο είναι το θέμα που δεν έχει συζητηθεί ακόμη εκτενώς, το θέμα των ε, διοικητικών πρακτικών των ε, επιχειρήσεων. Γιατί αυτό οι πρακτικές μιας επιχείρησης, οι πρακτικές της διοίκησης μιας επιχείρησης επηρεάζουν άμεσα την ευημερία των εργαζομένων στην επιχείρηση αυτή. Και όλα αυτά είναι απαιτητικά γιατί είναι δύσκολο μερικές φορέ για του πολιτικού ηθήνοντε για μας να αντιληφθούμε τι μέτρα χρειάζονται σε επίπεδο κυβέρνηση, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπής, για να βελτιωθούν οι διοικητικέ πρακτικέ των επιχειρήσεων, να αλλάξει ο τρόπο σκέψη, να έχουμε την κοινωνική καινοτομία. Και μάλιστα η επισκόπηση αυτή του Eurofound επιβεβαιώνει τι προκλήσει που εντοπίσαμε εμεί. Και χρήσιμο θα ήταν να έχουμε πρόσβαση και σε μια διεθνή συγκριτική ανάλυση. Γιατί γνωρίζουμε πολλά για την ποιότητα εργασία στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε την Ευρώπη με τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Και αυτό ίσως μας ε, οδηγεί σε ασφαλμένα συμπεράσματα πολιτικής. Γι' αυτό θα ήθελα να έχουμε μια επέκταση της επισκόπησης και σε άλλα μέρη του κόσμου. Θεωρείτε ότι έχουν γίνει αρκετά ώστε η ποιότητα στην εργασία να γίνει στόχος πολιτικής στην Ευρώπη. Ναι, είναι στόχος πολιτικής. Και σε όλα τα έγγραφα πολιτικής είναι στόχος φάμιλος με το στόχο για περισσότερες θέσεις εργασίας και καλύτερες θέσεις εργασίας. Και μάλιστα στα χθεσινά έγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική και από τη σημερινή φυσικά επισκόπηση στην Κυροφάν βλέπουμε ότι χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση αυτών των εγγράφων. Σίγουρα η πολιτική αυτή έχει συγκεντρώσει την προσοχή, αλλά δεν μεταφράστηκε σε ποσοτικούς στόχους, όπως το ποσοστό 75% απασχόλησης που γνωρίζουμε. Αλλά αυτό είναι αυτοαπόδεικτο. Αν δείτε την έκθεση, αν ακούσετε τις σημερινέ παρατηρήσεις και ομιλίες, διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει ένας δείκτης ή ένα ποσοστό που να αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε όλο το, όλη την αγορά εργασίας. Δεν είναι μονοδιάστατη διάστατη κατάσταση, υπάρχει μεγάλη πολυμορφία και δεν μπορούμε να συνοψίσουμε όλη την κατάσταση σε ένα ποσοστό, σε ένα νούμερο που να ισχύει για όλες τις ομάδες της εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Υπάρχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και όλα αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά χρήζουν διαφορετικές δράσεις, χρήζουν διαφορετικών δράσεων και φυσικά θα πρέπει να δούμε διάφορες πτυχές ε, των διαφόρων διαστάσεων. Δεν μπορούμε να τα συνοψίσουμε όλα σε ένα νούμερο ή ένα ποσοστό. Και Βέβαια το ότι δεν υπάρχει ποσοτικός, ποσοτικοποιημένος στόχος δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πολιτική που να προσανατολίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν λάθος να κάνουμε τέτοια απλοποίηση. Να, να περάσω στον κύριο Σκαρπέτα και να πούμε για τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρθηκαν για την ε, μέτρηση της ποιότητας. Εσείς πώς το επεξεργάζεστε. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να δώσω ουσιαστική απάντηση στη συζήτηση με αφορμή την ε, μελέτη των συνθήκων εργασίας. Βέβαια είμαι ένας ικανοποιημένος χρήστης της μελέτης και η συνεργασία μας ως τώρα υπήρξε ιδιαίτερα παραγωγική και στο πλαίσιο της ποιότητας ε, εργασίας. Ίσως καλό θα ήταν να επεκταθεί η μελέτη και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ξεκινήσω με ευχάριστα νέα το ξέρετε καλά εδώ, οι χώρες του G20 κάνουν λόγο για την ποιότητα εργασίας, για την εργασιακή ποιότητα. Από το 2015 έχουν υπόψη τους το στοιχείο αυτό ως κινητήρια δύναμη για καλύτερη ζωή των ατόμων και της κοινωνίας. Αυτό ίσως αν σας ακούγεται προφανές, αλλά αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι η συζήτηση για την ποιότητα γίνεται εδώ και καιρό και στο Eurofund και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον ΩΣΑ, αλλά πολλές φορές περιορίζεται. Περιορίζεται σε όσους ε, ε, ασχολούνται με θέματα της εργασιακής αγοράς. Νομίζω ότι η ποιότητα της εργασίας αυτή τη στιγμή έχει αναβαθμιστεί στην όλη συζήτηση των ε, πολιτικών ηγετών. Και το γεγονός ότι αυτό αυτή τη στιγμή αναφέρεται και στη δήλωση των, υπουργών, των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των G20 είναι ήδη ένα σημαντικό βήμα. Εάν μου επιτρέψετε και μια μια παρέκβαση. Ένα από του λόγου όπου δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα εργασία είναι και η διάρκεια αυτή του επαγγελματικού βίου. Υπάρχουν πολλά άλλα βέβαια σημάδια που οδηγούν προ τα εκεί, αλλά επειδή ανησυχούμε για την ποιότητα τη δουλειά, επειδή είναι πολύ πιο ε, εκτεταμένη η διάρκεια, προηγουμένω κοιτάζαμε περισσότερο τα ε, μισθολογικά, τι αμοιβέ, τι αποδοχέ κτλ. Τώρα βρισκόμαστε κάπου στο μέσο και η Υπουργοί Εργασία μιλάνε κάπω για το μέσο διάστημα μεταξύ τη δημιουργία θέσεων εργασία υψηλών προσόντων από τη μια και από την άλλη την ε, βάση τη όλη κατανομή. Πρέπει λοιπόν να δούμε το αποτέλεσμα που δίνει αυτό το μέσο διάστημα. Αυτό το μέσο διάστημα είναι που δημιουργεί το μέσο όρο. Το ενδιάμεσο επίπεδο δεξιοτήτων και τι ενδιάμεσε θέσει εργασία. Ο λόγο, και δεν θέλω τώρα εδώ να ε, εικάζω πάρα πολύ. Αυτό αποσχολεί του ε, πολιτικού ευθύνοντε, διότι αν κανεί διαβρώσει την μέση τάξη, διαβρώνει και το μέσο ψηφοφόρο. Και τελικά στι εκλογέ οι μέσοι ψηφοφόροι είναι αυτοί που αποφασίζουν. Ε, κλείνω την παρέκταση. Αυτό είναι ένα βήμα πρόοδου στο G20, το οποίο ακριβώς οφείλεται σε όλους τους φορείς που βρίσκονται εδώ και που έχουν εργαστεί τόσο σκληρά για το θέμα αυτό επί τόσο καιρό. Όμως η δουλειά η δική μας, του ILO, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής για την ε, Ευρώπη, και τη ΕΜΚΟ έχουν να κάνουν με όλα αυτά. Τι έχουμε κάνει στον ΩΣΑ τώρα. Ε, είναι θεμελιώδη σημασία να προσπαθήσουμε να έχουμε δείκτες οι οποίοι να είναι συγκρίσιμοι στον χρόνο μεταξύ των χωρών και στο μέγιστο δυνατό βαθμό να μπορούν να συνδεθούν με τις πολιτικές που χαράζουν οι θεσμοί. Αυτά στα πλαίσια της φιλοσοφίας μας για την ποιότητα της εργασίας. Με χαρά μου να πω ότι η συνεργασία μας ε, με τους συναδέλφους του ΑΕΛΟ έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο πλαίσιο, το οποίο το γνωρίζετε πολύ εδώ και το οποίο εγκρίθηκε από τον G20 Ω τρόπο για να δούμε πώ αναπτύσσεται και εξελίσσεται η αγορά εργασία. Και οι υπουργοί εκεί έθεσαν μια σειρά από πολιτικέ προτεραιότητε για το πώ να ε, προωθηθεί η καλύτερη ποιότητα τη εργασία. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, ε, μερικά από τα βασικά στοιχεία αυτού του πλαισίου που αναπτύξαμε. Τρει διαστάσει. Πρώτα απ' όλα η ποιότητα των εισοδημάτων. Δεν μιλάμε για την έλλειψη εισοδημάτων, που βεβαίω είναι κάτι το πολύ σημαντικό όπω είπε η Μανουέλα, για την καλή διαβίωση των ατόμων, αλλά και η κατανομή των εισοδημάτων. Και αυτό έχει σημασία για το πώς οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ολοκληρώνονται καθώ δουλεύουν σε μια ελεύθερη αγορά εργασία. Κοιτάζουμε την ασφάλεια. Ο κίνδυνο να χάσει κανεί τη δουλειά του για διαφορετικού ε, λόγου. Αλλά και το τι παίρνει ο καθένα εφόσον χάσει τη δουλειά του. Και βεβαίω από τη μελέτη των ε, θετικών εργασία βλέπουμε και το εργασιακό περιβάλλον. Αυτό το δείκτη τον χρησιμοποιούμε για να αξιοποιήσουμε και τα μακροοικονομικά στοιχεία που έχουμε, όχι μόνο με υποκειμενικά αλλά και με αντικειμενικά στοιχεία. Έχουμε δηλαδή μια έννοια αλυσίδα θέσεων εργασία. Το τι κάνουν οι άνθρωποι στη δουλειά τους, πώ αισθάνονται γι' αυτό, αλλά και πώς το αξιοποιούν. Δηλαδή, εάν κανείς ε, είναι σε μια θέση που έχει τη συγκεκριμένη πίεση και τις συγκεκριμένε απαιτήσει, βρίσκεται σε μια χαμηλότερη θέση. Αυτό το τμήμα ε, τροφοδοτεί και εμπλουτίζει τη στατική μας για την εργασία, αλλά στις ε, οικονομικές επισκοπήσεις ένα χώρα χρησιμοποιούμε το στοιχείο της εργασίας για να δούμε τι πολιτικές πρέπει να σχεδιάσει κάθε χώρα επιμέρους. Οι τρεις διαστάσεις δεν σας ε, εκπλήσει. Αν δει κανείς αυτά που είπαμε, αμοιβές, ε, κατανομή μισθολογικά, είναι γνωστά από καιρό. Αυτό που είναι καινούριο είναι η ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Να υπογραμμίσω αυτό πώς επηρεάζει τη δική μας την προσέγγιση. Να πάω πίσω σε αυτό που είπε και ο Τόμ. Δεν είναι ο λόγο ότι απλώ καταλάβαμε ότι η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντο είναι καθοριστική για την εργασία, αλλά υπάρχει και όλο ένα και περισσότερη βιβλιογραφία που δείχνει ότι η καλύτερη ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον είναι καλή και για την παραγωγικότητα. Πολλή δουλειά γίνεται στην επισκόπηση τη απασχόληση για να δούμε το ποιε είναι οι πρακτικέ εργασίε που έχουν υψηλέ αποδόσεις. Οι εταιρείε που τι εφαρμόζουν όχι μόνο έχουν καλύτερε εργασιακέ συνθήκε για του εργαζομένου, αλλά έχουν και καλύτερα, καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και μεσοπρόθεσμα με δυναμικό για ανάπτυξη. Άρα η ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντο, τι δικέ μα αναλύσει, ξεπερνά λιγάκι την απλή αποτίμηση του πώ αυτό επηρεάζει την ε, ευεξία των ίδιων των εργαζομένων. Αλλά μα απασχολούν και τα μακροοικονομικά στοιχεία τη αγορά. Μιλήσατε για κατευθυντήριε γραμμέ. Έχουμε αυτή την υπέροχη μελέτη κάθε πέντε χρόνια, η οποία ισχύει μόνο για χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητήσαμε τη δυνατότητα να επεκταθεί γεωγραφικά. Σε συνεργασία με τον Eurofund. Το είπε και ο Όσα. Όμω χρειάζονται πληροφορίε πιο συστηματικά. Δηλαδή αυτό που κάνουμε με τι κατευθυντήρε γραμμέ που σχεδιάζουμε με του συναδέλφου των στατιστικολογικών υπηρεσιών είναι να δούμε πού τα βασικά σημεία, όσων περιλαμβάνει η έκθεση του Φαν, μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλε υπάρχουσε μελέτε έτσι ώστε να δίνουν πιο συχνά στοιχεία για να μπορούμε να μετρώμε ε, πώ εξελίσσεται η αγορά εργασία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στατιστικολόγοι μα, όχι μόνο των ευρωπαϊκών χωρών, όλων των χωρών του ΩΣΑ, δραστηριοποιούνται εδώ και θέλουμε να ξεπεράσουμε και, άλλα, και τα όρια του ΩΣΑ ενδεχομένω, γιατί και κάποιε αναδυόμενε οικονομίε συνεργάζονται μαζί μα. Του προσφέρουμε διαφορετικέ επιλογέ. Τρει βασικέ επιλογέ. Πρώτον, μια εκτεταμένη μελέτη με συγκεκριμένα έντυπα που καλύπτει τι βασικέ διαστάσει που μα επιτρέπουν να ορίσουμε καλύτερα την ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Ε, μια συμπυκνωμένη μελέτη, λιγότερο φιλόδοξη, αλλά συμπεριλαμβάνει τι βασικέ ε, παραμέτρου που χρησιμοποιούμε στην ε, έτσι καλλιώ ε, κεντρική μα μελέτη. Και μετά την πιο απλή που μπορεί να εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα, ε, ένα ερωτηματολόγιο πολύ απλό, πολύ απλοποιημένο, με κάποιε βασικέ ερωτήσει. Ε, αλλά αν θέλουμε να δούμε τα βασικά στοιχεία ε, όλων των μελετών μαζί, εκεί μπορεί κανεί να μελετήσει τι προποθέσει, του όρου τη αγορά εργασία και την ποιότητα κατά επέκταση. Νομίζω λοιπόν ότι αν η ποιότητα τη αγορά εργασία βρεθεί στο επίκεντρο τη προσοχή των πολιτικών εθνών και εφόσον τώρα μετρούμε τη σχετική πρόοδο με την ποιότητα, την εργασιακή ποιότητα, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και συστηματικά δεδομένα, όχι μόνο κάθε πέντε χρόνια. Σε ένα βαθμό αυτέ είναι οι προκλήσει μα και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτή είναι η συνεισφορά μα από τον ΩΣΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ σαφέ. Σαφέ. Λοιπόν, πάμε τώρα ε, από τον δικό σα τομέα στον κόσμο ολόκληρο, στον Διεθνή Οργανισμό εργασία. Θα ήθελα λοιπόν να μα πείτε τι σημασία έχουν οι συνθήκε εργασία στον ILO και να σας πω κάτι, είχαμε ενημερωθεί τότε πως η έρευνα αυτή για τις συνθήκες εργασίας χρησιμοποιούνταν ακόμα και σε χώρες όπως η Τανζανία και μας εξηγήσατε ακριβώς ποια ήταν η χρήση που γινόταν. Μπορείτε λίγο να μας εξηγήσετε περισσότερα πράγματα και την πολιτική τους χρήση. Αν μου επιτρέπετε, πριν αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο είπε ο Στέφανο, γιατί πράγματι παρά την διάβρωση, θα έλεγα, της ποιότητας εργασίας παντού στον κόσμο, το θέμα της ε, ποιότητας δουλειάς είναι θέμα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους G20 και στον ΑΕΛΟ. Αλλά αυτό το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι υπάρχει ατζέντα του 2030 για την αηφόρο ανάπτυξη που πράγματι αποδίδει μεγάλη σημασία στο να επερλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι μέσω της αξιοπρεπούς εργασίας και της παραγωγικής και ακριβώ τώρα που προσπαθούμε να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογή και την κάλυψη των ευρωπαϊκών αυτών ερευνών σε άλλα μέρη του κόσμου. Και βεβαίως ε, υπάρχει μεγαλύτερη διάθεση να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού και να γνωρίζουν όλοι ότι οι ποιοτικέ θέσει εργασία έχουν μεγάλη σημασία ακριβώς για κοινωνίες με περισσότερη συμπεριλήψη και αυτό που σωθούν όλοι μας οι οργανισμοί. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω την σημασία των εμπειρικών δεδομένων για το γεγονός πως οι ποιοτικές θέσεις εργασίας είναι καλές για την παραγωγικότητα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και βεβαίως όλοι το αντιλαμβανόμαστε, είναι προφανές. Και βεβαίω σημασία έχει και να το αποδεικνύουμε, γι' αυτό θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ στις προσπάθειες που γίνονται στον ILO για να καταγραφεί και να αξιολογηθεί η σχέση μεταξύ της βελτίωσης των ε, συνθήκων εργασίας με την παραγωγικότητα. Γιατί κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει πολλές πολλές συζητήσεις είναι το αν η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι προαπαιτούμενο για το εάν θα έχουμε καλύτερες ε, περισσότερες ε, και παραγωγικότερες δουλειές ή με το να επενδύσουμε στις συνθήκες εργασίας θα έχουμε μεγαλύτερη παραγωγικότητα που είναι η άλλη σχολή σκέψης και βέβαια προσπαθούμε και εμείς ακριβώς να δούμε αυτή την προσπάθεια σε ολόκληρη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα σε χώρες που, είναι, που παράγουν τα εμβήματα για την αγορά των ΙΠΑ στις οποίες ο ΑΙΟΛΟ εργάζεται 10 χρόνια για να βελτιώσει ακριβώς ε, τις συνθήκες εργασίας μέσω της ε, μεγαλύτερης συμμόρφωσης. Και τα στοιχεία είναι πραγματικά συγκλονιστικά υπάρχει μια σαφής αιτιώδης ε, σχέση μεταξύ βελτίωσης των ε, συνδικών εργασίας και της παραγωγικότητας. Τώρα, για το πώς προσπαθούμε να δούμε αυτά τα ζητήματα σε χώρες όπου η αγορά εργασίας έχει μεγάλη ανεπίσημη απασχόληση και άρα ίσως υπάρχει ένα λιγότερο ενδιαφέρον για μια τέτοια ανάλυση ή βελτίωση των συνθήκων εργασίας. Οφείλω να πω ότι πράγματι ε, λειτουργεί κάτι τέτοιο, ειδικά σε χώρες μέσου εισοδήματος και χαμηλού. που εμπορεύονται εξαρτή με αυτό το μέρος του κόσμου. Οι οποίες ε, τα τελευταία έτη λόγω της αύξησης των τιμών των ε, αγαθών λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επίσημων θέσεων εργασίας καταφέραν να μειώσουν τις ανισότητες με το να επενδύσουν σε τέτοια θεσμικά όργανα της αγοράς εργασίας όπως η Κίνα, η Βραζιλία και η Αργεντινή πριν ε, την ύφεση των τελευταίων ετών. Όταν βελτιωνόταν λοιπόν η οικονομική κατάσταση ήθελαν βεβαίως και οι χώρε να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας για να δημιουργηθεί και μια εγχώρια ζήτηση και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε εξαγωγές για να αναπτυχθούν. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ και βεβαίως περνάμε τώρα στις ερωτήσεις. Από την Παρακαλώ εσείς να ακούσουμε τρεις ερωτήσεις και μετά απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Λέω από το ΣΕΝΕΡΕΣ για το συγκριτικό δίκαιο του εργασιακού, της εργασιακής νομοθεσίας και της ασφάλειας στην εργασία από το Πανεπιστήμιο του Μπορντό. Η μελέτη του Eurofond ε, εντάσσεται σε ένα νομοθετικό πλαίσιο κοινοτικό με την οδηγία πλαίσιο της 12 Ιουνίου του 1999, τις οδηγίες και κείμενα για την ασφάλεια και την υγεία στην αγορά εργασία, την οδηγία για την καταπολέμηση των διακριτικών μεταχειρήσεων, υπέρ της ισότητας ανδρών γυναικών επίσης. Είναι σημαντική αυτή η βοήθεια που δείχνει ότι τα κοινοτικά κείμενα μεταφέρονται στην νομοθεσία ε, βάσει του πνεύματος, των στόχων και των συνεπειών που επιδιώκουν. Και βλέπουμε κιόλα αν υπάρχει πραγματική αλλαγή στι εθνικέ πολιτικέ. Τώρα, χρειάζεται ένα νέο κείμενο. Τέθηκε το ερώτημα και προηγουμένω. Όχι, γιατί κάποια ενδιαφέροντα και εύστοχα κείμενα υπάρχουν και απλώ πρέπει σωστά να υλοποιηθούν. Η απάντηση λοιπόν για την αποτελεσματικότητα των κειμένων των νομοθετημάτων είναι το κατά πόσον σωστά μεταφέρονται και υλοποιούνται. Έτσι κι αλλιώς το πόρισμα της μελέτης μας ε, υποχρεώνει να φροντίσουμε να καταργήσουμε τα όρια και τα σύνορα μεταξύ των συνομιλητών και να αλλάξουμε μοντέλο. Από το μοντέλο της ε, ε, διόρθωσης να περάσουμε στο μοντέλο της πρόληψης, να ασχοληθούμε και με την εργασία και όχι μόνο με την έλλειψή της και να δημιουργήσουμε ίσως γέφυρες μεταξύ των οικονομικών συλλογισμών και της υγείας στην εργασία. Με, άλλη, με άλλα λόγια, μήπως είναι δυνατόν, μήπως μπορούμε να σκεφτούμε μια νέα προσέγγιση του ορισμού της οικονομίας, μια νέα οικονομία που να συμπεριλαμβάνει την υγεία στην εργασία έτσι ώστε να συνδυάσει την υγεία από τη μια με την παραγωγικότητα από την άλλη επιτρέποντας να, να δηθούν παιδεία καινοτομία και καινοτομίε τέτοιε που να λαμβάνουν υπόψη του την υγεία των εργαζομένων με σκοπό να αλλάξουν οι συμπεριφορέ. Όλοι θα είχαν ωφεληθούν από αυτό και ολοκληρώνοντα πρέπει όλοι οι φορεί, κοινωνικονομικοί, πολιτικοί να εμπλακούν. Ευχαριστώ, αλλά και άλλοι ζήτησαν το λόγο. Κρίς μίστερ από την Ένωση Εργαζομένων του Βελγίου. Θα είμαι κάπως ομός, ο συνήθως, μάλλον. Το δικό μου το συμπέρασμα είναι ότι από το πολιτικό και επίπεδο στρατηγική, στρατηγικού σχεδιασμού δεν έχουμε πολλά να περιμένουμε. Ακούσαμε ένα σωρό ανθρώπου να περιγράφουν ότι υπάρχουν διαφορετικέ διαστάσει και πολλέ ε, παράμετροι που παίζουν ρόλο. Κάποιες είναι έμφυτες, κάποιες είναι εξωτερικές από το αντικείμενο της εργασίας, δηλαδή τι θεωρεί κανείς ουσιαστικό, τι θεωρεί σκόπιμο και απάντηση ξαφνικά είναι ρύθμιση. Εδώ η έκθεση μας είπε ότι δεν υπάρχει κάτι που να είναι λύση για όλα και ενός μεγέθους. Δεν υπάρχει one size fits all. Και η απάντησή σας είναι ρύθμιση. Πώς γίνεται. Μιλάμε για συντελεστές σε Τομεί που οι συντελεστέ είναι τελείω αντικειμενικοί και μετρήσιμοι, πάλι δεν είναι ξεκάθαροι δείκτε. Πρέπει να υπάρχουν συγκρίσιμοι δείκτε. Πώ θα γίνει αυτό σε αυτό το τομέα. Σε 20 χρόνια ακόμα δεν θα έχουμε τίποτα, εάν έτσι προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την έννοια του burnout. Μιλάμε για ανθρώπου που έχουν χάσει το κίνητρό του για τη δουλειά. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σε καταστάσει και σε φορεί όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα χρυσό κλουβί Φανταστικέ αμοιβέ, δεν έχουν όμω προκλήσει. δεν βρίσκουν ε, ότι έχει κανένα σκοπό, κανένα νόημα η δουλειά του. Αυτό συμβαίνει και στα θεσμικά όργανα και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Μήπω αυτό να κοιτάξετε και μετά να ξανάρθετε να μα τα πείτε, αν βρείτε τι σωστέ απαντήσει, την προσέγγιση, αυτή η ποιότητα εργασία να αυξηθεί. Η απάντησή μου είναι θα πρέπει να εργαστούμε στο χώρο εργασία, τον ίδιο, με του εργαζομένου, με του μεσαίου μάνατζερ, και με εξωτερικούς ε, ειδικού ενδεχομένους. Να δούμε την ποιότητα ακριβώ στο ίδιο το χώρο που εργάζονται οι άνθρωποι, την προσωπική κατάσταση του καθενό. και εκεί να προσπαθήσουμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ των φιλοδοξιών του, των ικανοτήτων του και την κατάσταση τη δουλειά του. Να του δώσουμε δυνατότητε, να συνεχίσουν να καλλιεργούν τι δεξιότητέ του, να είναι απασχολήσιμοι καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα. Συμφωνείτε καθόλου με αυτό? πρόκληση η ερώτησή σας, αλλά να τη θέσουμε στου πανελίστ. Και μια τρίτη ερώτηση για τον γύρο αυτό. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση, λίγο γενική μάλλον, κυρίως για τον κύριο Σκαρπέτα, αλλά και για τους υπόλοιπους πανελίστ. Ο κύριος ε, Σκαρπέτα είπε ότι υπάρχει υποβάθμιση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και αναφέρατε και το πρόβλημα των ενδιάμεσων θέσεων εργασία, το οποίο αρχίζει να γίνεται προεξάρχων. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το εξή. Τι άποψη έχετε για τη συνοπτική εικόνα αυτών των ενδιάμεσων θέσεων εργασία στο πλαίσιο των γιγαντοοικονομιών και την ταχύτατη ατάκιστη θα έλεγα ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του κόσμου μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο προς τον Τόμ για την πρώτη ερώτηση, για την αλλαγή του τρόπου σκέψη που πρέπει να εφαρμόσουμε πρώτα απ' όλα. Καθόλου εύκολη. Οι δύο πρώτες ερωτήσεις ε, περιέχουν το ίδιο μήνυμα. Νομοθεσία και ρύθμιση που αφορούν την ποιότητα, την υγεία, στο χώρο εργασίας θα πρέπει να επικαιροποιηθούν γιατί συνήθως κανονισμούς έχουμε αλλά αυτοί δεν πρόκειται να αλλάξουν. Το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το συνολικό πλαίσιο πολιτικής και πώς εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσουμε τις εμφανείς απειλές που βλέπουμε, τις αβεβαιότητες, τη ραγδαία τεχνολογική αλλαγή, δημογραφικές αλλαγές, την παγκοσμιοποίηση και το μάλλον αβέβαιο πολιτικό κλίμα που επικρατεί. Πώς θα αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις, διαφυλάσσοντας την ανταγωνιστικότητά μας και ταυτόχρονα και το κοινωνικό μας μοντέλο. Και αυτή σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση από τη συζήτηση για τους κανονισμούς, τις ε, ρυθμίσεις και τις νομοθετικές διατάξεις. Αυτό βέβαια το λέει κάποιος που ο ρόλος του είναι να προεδρεύει σε μια επιτροπή που ασχολείται με μείζονες επιλογές στρατηγικής και νομοθεσία. Δεν θα έπρεπε να το λέει αυτό ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που επίσης έχει τέτοιο νομοθετικό και νομοπαρασκευαστικό ρόλο. Αλλά ίσως αυτός είναι και ο συνδετικός κρίκος για να απαντήσω και στην ε, ερώτηση του Κρίς. Όντως, αν δεν περιμένεις από τους πολιτικούς ηθήνοντες να λύσουν τα προβλήματα, εμείς περιμένουμε πραγματικά από τους κοινωνικούς εταίρους στον χώρο εργασίας να λύσουν τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν η κυρία Τομέη θα ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση αν όντως χρειαζόμαστε περαιτέρω κανονιστική ρύθμιση και αν θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρος τις περαιτέρω ρυθμίσεις και να επικεντρωθούμε στο θέμα της εργασίας και της ποιότητας. Σίγουρα μια αποκλειστική εστίαση στην κανονιστική ρύθμιση είναι ανεπαρκής. Και επανέρχομαι εδώ στο σχόλιο του Κρίς. Βέβαια χρειάζεται και η κανονιστική ρύθμιση, γιατί καθορίζει με σαφήνεια τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ε, ενθαρρύνει κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά και στον τρόπο σκέψης, προκειμένου να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες. Μερικές φορές η πρόκληση μπορεί να μην είναι η θέσπιση νέων νομοθετικών διατάξεων, αλλά περισσότερη εφαρμογή των ε, ισχυουσών διατάξεων. Και ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε τι μείγμα κινήτρων και φοβήτρων ή κυρώσεων θα ενίσχυαν το βαθμό συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Και σίγουρα η βελτίωση της συμμόρφωσης με την νομοθεσία ε, βελτιώνει τις εργασιακές συνθήκες και ενισχύει και την παραγωγικότητα. Και οι επιχειρήσεις που δείχνουν πρόοδο από αυτή την άποψη λαμβάνουν και κίνητρα με τη μορφή ε, μεγαλύτερης πρόσβασης σε συγκεκριμένες αγορές. Του τουλεχθέντος, ε, αυτό ήταν και ένα θέμα που έδειξε το πρωί ο Μισελ Σαββό. Είπε λοιπόν ότι υπό το φως των αλλαγών ε, των ε, μεταρρυθμίσεων, των μετασχηματισμών που γίνονται, στη φύση της εργασίας, ε, στις εργασιακές ρυθμίσεις που απάδουν από τις παραδοσιακές ε, εργασιακές σχέσεις, δημιουργούν πολλές νέες προκλήσεις. Για παράδειγμα, η διασφάλιση της κοινωνικής προστασίας. Οπότε ρώτησε, χρειαζόμαστε άλλους κανονισμούς ή είναι κατάλληλη η ισχύοντες κανονισμοί. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσουμε. Και όταν ε, μιλούμε για τις ε, gig economy, shade economy, την αλληλεξάρτηση των θέσεων απασχόλησης, μερικές φορές οι διαχωριστικές γραμμές είναι πολύ ρευστές και πολύ ανεξάρτητοι αυτοαπασχολούμενοι που ναι με χαρακτηρίζονται αυτοαπασχολούμενοι ανεξάρτητοι αλλά παρόλα αυτά ε, βρίσκονται σε μια θέση εξάρτησης ενώ δεν τη χάνουν της προστασίας. Ίσως ε, η ερμηνεία της εργασιακής σχέσης δεν είναι αρκετά ευρεία ώστε να καλύπτει τις μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στον εργασιακό κόσμο. Οπότε η κανονιστική ρυθμίση είναι έτοιμα της συζήτηση. Ναι, σε ό,τι αφορά τις ε, ε προοπτικές αυτών των ε, μεσαίων ε, διάμεσων θέσεων και αν υπάρχει ανάγκη επίσης για περισσότερη νομοθεσία, περισσότερη κανονιστική ρύθμιση. Σίγουρα θέλουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα των θέσεων εργασία και η λύση είναι κανονιστικές ρυθμίσεις, αλλά ίσως θέλουμε καλύτερες κανονιστικές ρυθμίσεις και φυσικά να λαμβάνουμε μέρος στη συζήτηση αλλά θα πρέπει επίση να εξετάσουμε το θέμα τη εφαρμογή, το βαθμό εφαρμογή τη ισχύουσα νομοθεσία. Και αυτό που κάνουμε και στον ΩΣΑ είναι να δούμε ε, τι αποτελέσματα έχουν για διάφορες ομάδες εργασίας ε, οι καταστάσεις στην αγορά εργασίας. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα που βλέπουμε σε διάφορες ομάδες εργαζομένων, κρίνουμε αν είναι κατάλληλη η νομοθεσία, χρειάζεται επιπλέον νομοθεσία και τι χρειάζεται για να βελτιωθούν οι εργασιακές συνθήκες. Προσοχή λοιπόν. Αλλά σας ευχαριστώ που διευρύνατε κάπως τη συζήτηση και είπατε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε την ε, πρωταρχική μας, ε, τον πρωταρχικό μας προσανατολισμό και αν είναι ε, η παραγωγικότητα το ζητούμενο. Ίσως θα πρέπει να, από την παραγωγικότητα να περάσουμε περισσότερο σε έναν σε μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και εδώ η ποιότητα της εργασίας μετράει. Και επίσης η πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση. Και σίγουρα σε αυτά τα σημεία κάπως χωλαίνομαι. Και είναι η δεύτερη φορά που οι χώρες του G20 λένε ότι θέλουν να προωθήσουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Και εμείς προσπαθούμε στην ομάδα εργασία να δημιουργήσουμε τις βάσεις για να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι αφορά την ερώτηση του Κρίς, Συνεχίζω του προλαλήσαντε και θεωρώ ότι περισσότερε δράσει θα πρέπει να ληφθούν στον χώρο εργασία. Οπότε ο διάλογο μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων είναι εδώ ζωτική σημασία. Ο ρόλο τη πολιτική είναι σημαντικό μεν, αλλά ανεπαρκή δε. Και στον ΩΣΑ έχουμε την ασφάλεια την ανασφάλεια του χώρου εργασία, που είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει να προλάβουμε πιθανέ διαρθρωτικέ αλλαγέ και να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις να προλάβουν τις αλλαγές και να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να προσαρμοστούν σε αυτές τις αλλαγές. Παρόλο που μερικές φορές αλλαγές προϋποθέτουν και απολύσεις και ανάγκη ανέβρεση νέες θέσεις απασχόλησης. Πάντως η πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο και κάναμε μια αξιολόγηση και είχαμε πολλά καλά παραδείγματα του τι πολιτική χρειάζεται για να βελτιώσει την κατάσταση και να έχουμε υψηλές εργασιακές, υψηλής απόδοσης εργασιακές πρακτικές και από αυτήν την άποψη χρειαζόμαστε και πολιτική. Τώρα, οι προοπτικές, εδώ δεν είναι θέμα μόνο ανεξάρτητης εργασίας σχέση με την gig economy. Εδώ περισσότερο μιλούμε για τις μισθωτές εργασίες. Πάντως οι προκλήσεις είναι να βοηθήσουν αυτού που θα αλλάξουν τον τρόπο δουλειά του, να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα που χρειάζονται, είτε να κρατήσουν τη θέση εργασίας τους, είτε να βρουν εύκολα άλλη θέση εργασίας. Ε, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να εμπλουτίσουν ίσως τα προσόντα και τις δεξιότητες τους. Για να πούμε δύο λόγια, δηλαδή, λοιπόν, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τι πολιτικέ μα για τη διαβίου κατάρτιση, γιατί Πουθενά στην Ευρώπη ο άλλου δεν είμαστε επιτυχείς αυτό. Και εκεί οι εργοδότες θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για την συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων σε μια οικονομία που μεταβάλλεται για να αναλάβουν και καθήκοντα που απαιτούν νέε δεξιότητες και προσόντα. Ψηφιακή οικονομία, νέε μορφέ ανεξάρτητη εργασία. Θα πρέπει να δούμε πρώτα τα στοιχεία. Αυτό το έργο ήδη καλύπτεται από τα ισχύοντα συστήματα κοινωνική προστασία. Όχι, μάλλον σίγουρα όχι σε, στον ίδιο βαθμό για όλους τους ε, εργαζόμενους. Οπότε μια κοινωνική προστασία μπορεί να είναι πιο περιεκτική, πιο γενική, ώστε να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, άσχετα με το είδο σύμβαση που έχουν. Βέβαια, είναι πολύ απαιτητικό αυτό το πρόγραμμα, να κάνουμε ένα απολογισμό της παρούσας κατάστασης, να δούμε το έβρος της κάλυψης, ίσως να το παρατείνουμε περαιτέρω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και επίσης να εξοπλίσουμε τους εργαζομένους με προσόντα, με εφόδια, γιατί η προστασία θα πρέπει να είναι για τον εργαζόμενο, όχι για την σύμβαση. Γιατί πολλοί εργαζόμενοι κάνουν δύο και τρεις δουλειέ ταυτόχρονα. Οπότε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κοινωνική προστασία στον εργαζόμενο και το δικαίωμα στην κατάρτιση και τη δυνατότητα να επιλέξει την κατάρτισή του. Αυτή θα είναι σημαντική πρόκληση για το μέλλον. Μάλιστα. Κοιτάξτε, όχι και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον Κρίς εδώ, ότι πρόκειται για πράγματα που είναι στο επίπεδο των εταιριών. Δηλαδή πολλές από τις καλύτερες λύσεις θα βρεθούν στο επίπεδο της κάθε εταιρεία, όπου γνωρίζουν ακριβώς ε, τα δυνατά τους και τα ασθενή τους σημεία. Και είναι εύκολο να συμφωνήσουμε μαζί σας, γιατί και η έρευνα σας δίνει τα στοιχεία. και βεβαίως ε, το 1 τρίτο των εργαζόμενων που εργάζονται ε, σε οργανισμούς με χαμηλή διακριτική ευχέρεια ε, βλέπουμε ότι έχουν την αντίθετη άποψη από αυτούς που δουλεύουν σε οργανισμούς με υψηλότερη διακριτική ευχέρεια οι οποίοι μετά βεβαίως έχουν και καλύτερα αποτελέσματα, κάτι το οποίο βέβαια είναι και θετικότερο για τις ε, εταιρείε. Και μετά να δούμε μια άλλη έρευνα για τις εταιρείε. Έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Και εδώ πέρα μιλάμε για ε, εταιρείε, ε, την διοίκηση και τα υψηλά επίπεδα άμεσης και έμεσης συμμετοχής, κάτι το οποίο σημαίνει υψηλή ικανοποίηση των εργαζομένων και καλύτερη οικονομική απόδοση για την εταιρεία. Οπότε, τα στοιχεία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το ότι ε, εάν το 1 τρίτο των επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις χαμηλής εμπλοκής και δεν υπάρχει κάποια εκπροσώψη των εργαζομένων, εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο διάλογος αυτός πρέπει να ξεκινήσει από αυτά τα ζητήματα που είναι εύκολο νομίζω να συμφωνήσουμε ότι λύνονται στο επίπεδο της εταιρείας. Μάλιστα, έχουμε ακόμα χρόνο εγώ με τον Κρίς να συζητήσουμε το θέμα της ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων σε εταιρείε όπου δεν υπάρχει κοινωνικός διάλογος, αλλά αυτό είναι βελγική συζήτηση, ενδοβελγική. Έχουμε λίγο χρόνο για άλλες ερωτήσεις αν έχετε. Ναι, παρακαλώ εσείς. Κοιτάξτε. Μιλήσατε για τι ε, διάφορε υπηρεσίε απασχόληση στην Ευρώπη και τα διαφορετικά πρότυπα που ισχύουν. Ε, είδαμε όμω το χώρο εργασία να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία. Μιλήσαμε για οικονομία, μιλήσαμε για το χάσμα το μισθολογικό. Οι διεμηνεί δεν μπορούν να σα να σας καταλάβουν ακριβώ. Μπορείτε να μιλάτε ίσω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Θα, έχω μια, θα είχα μια ερώτηση για το θέμα των προτύπων και την απασχόληση. Δεν ξέρω αν αυτή η διαφοροποίηση είναι η πλέον εύστοχη. Διότι αυτό που βλέπουμε είναι η αγορά εργασία να γίνεται πολύ πιο ετερογενή και επικοινόμορφη. Έχω σοβαρέ αμφιβολίε για το κατά πόσον είναι σκόπιμη η διάκριση τη χαμηλή και ψηλή ποιότητα. Βλέπουμε στην πραγματικότητα, εάν δούμε το τι συμβαίνει, οι εταιρείε και επιχειρήσει να προσφέρουν κάποιες λύσεις, να προσπαθούν να γίνουν πιο καινοτόμε με ωφέλη που όμως δεν ε, έρχονται πίσω στους ίδιους τους εργαζομένους. Αυτό ισχύει σε πολλές χώρες. Γι' αυτό λοιπόν να σκεφτούμε συστήματα ασφάλισης καινούργια καινοτόμα και τις πάγιες ή μη πάγιες πρακτικές μας. Έπειτα, ένα επιπλέον σημείο για το μέλλον της αγοράς εργασίας και από τόπου στο διαδίκτυο, όταν κοιτάζουμε τα στοιχεία, να δούμε και αυτά που έχουν πρόσφατα δημοσιευτεί. Oui, Ένα τελευταίο ε, σχόλιο από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία εργασία. Από το πρωί μιλάμε για την ποιότητα της εργασίας. Εδώ δεν έχουμε αναγκαστικά την ε, πιο ε, εύστοχη προσέγγιση. Πολλά υπόθηκαν για τη διοργάνωση της εργασίας, για αυτό που είναι κεντρική σημασία. Δηλαδή ο εργαζόμενος ε, παρεμβαίνει στην εργασία του και καθορίζει την ποιότητά του. Ο οργανισμός, η διοργάνωση μάλλον, στο εργαστήριο, στην επιχείρηση, στο συνεργείο ε, καθορίζεται από τον ίδιο τον, τον εργαζόμενο. Και ακούσαμε και κάτι άλλο να λέγεται πολύ το χάσμα μεταξύ όσων έχουν πολύ καλές συνθήκες εργασίας και όσων έχουν πολύ δύσκολες. Η ψαλίδα είναι τεράστια, απίθμενη. Το χάσμα αυτό λοιπόν είναι τεράστιο. Βλέπουμε ότι η επισφαλής εργασία, η προσωρινή μάλλον εργασία ήταν η πόρτα από την οποία αφήσαμε να εισχωρήσει και να διεισδύσει η επισφάλεια στην αγορά εργασίας. Εκπλήσουμε που σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε επιχείρηση που μπορεί να παρεμβαίνει και έχει διωχθεί για δήλωτη εργασία. Εμένα αυτό πραγματικά με σοκάρει. Έτσι, η κατασκευαστική εταιρεία, λέω. Μεγάλη κατασκευαστική γαλλική, η οποία έχει και κανάλι τηλεοπτικό στη στην κατοχή τη και το καθεξής. Διώχθηκε ε, για δήλωτη εργασία, για προσωρινή εργασία που στην ουσία ήταν αδήλωτη δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι ένας εργαζόμενος θα έχει όλα τα προνόμια και τα δικαιώματα και ο άλλος κανένα. Και θα πρέπει να ικανοποιείται με ό,τι του δίνουμε. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Βρείτε μια ισορροπία μεταξύ των δύο. Η σχετική νομοθεσία υπάρχει. Και νομίζω το ξέρετε κι εσείς πάνω από 20 χρόνια. Είμαι στατευμένο εγώ και τα γνωρίζω. Η νομοθεσία δεν είναι κάτι που δεν εφαρμόζουν συνήθω οι μικρέ επιχειρήσεις. Οι μεγάλε λιγάκι την παρακάμπτουν και την προσαρμόζουν στι ανάγκες του. Αυτά. Μπάρμπαρα. Ήταν ε, παραδρομή όταν είπε κάτι αρνητικό για τις ε, ε, από τα γραφεία βρέσεως προσωρινής εργασίας. Ε, υπενήχθηκες κακή εργασιακή ποιότητα. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει η έκθεση, η μελέτη, είναι ότι το καθεστώς του εργαζομένου, της εργασίας μάλλον, έχει σημασία για την εργασιακή ποιότητα. Και βλέπουμε αφένα στους αυτοαπασχολούμενους ε, και τους ε, μισθωτούς ε, με συμβάσεις αορίστου έχουν κατά μέσο όρο καλύτερα αποτελέσματα σε αυτούς τους δείκτες εργασιακής ποιότητας από όσους έχουν προσωρινές ή ε, περιορισμένου χρόνου συμβάσεις εργασίας ή αυτούς που είναι ψευτό αυτοαπασχολούμενοι. Αυτά είναι τα αποτελέσματα υψηλού επίπεδου και ήδη από το χρόνο θα ξεκινήσουμε μια δευτερογενή ειδική ανάλυση για αυτή τη σχέση μεταξύ του ε, καθεστώτος απασχόλησης και των εργασιακών συνθήκων. Πάντω συμφωνώ μαζί σα ότι χρειάζεται πιο εμπεριστατωμένη και εντελεχέστερη ανάλυση για το πώ διάφορες μορφές μη ε, χαρακτηριστικής τυπικής εργασίας επηρεάζουν τις εργασιακέ συνθήκες. Ευχαριστώ. Ο Τόμισο, ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι ε, δεν είναι εύκολο να κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ τυπικών και μη τυπικών ε, μορφών εργασίας και σίγουρα οι εργασιακές ε, σχέσεις γίνονται όλο και πιο πολύμορφες και αναμοιόμορφες και καλύτερα να επικεντρωνόμαστε περισσότερους στους ανθρώπους, στους εργαζόμενους και όχι στις συμβάσεις και να δούμε τι γίνεται σε επιχειρήσεις, σε τι πρακτικές εφαρμόζουν. Γιατί υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν κάποιες καλές θέσεις εργασίες ε, από ε, γραφεία, και καλές αποσπάσεις και φαντάζομαι και μερικοί από εσάς εδώ είστε αποσπασμένοι, μερικοί ίσως και στη Eurofound, στο Ίδρυμα Eurofound. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν και αυτές τις διαφορές. Να μην κατηγορηποιούμε τους ανθρώπους ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν. Και αυτήν την άποψη η επισκόπηση μας βοηθά να στηρίξουμε την ανάλυση μας στα πραγματικά βιώματα των εργαζομένων για τις εργασιακές τους συνθήκες και όχι να τους κατηγοριοποιούμε σε ευρύτατες ε, διοικητικές κατηγορίες. Είμαστε κατά τέτοιου διαχωρισμού αυτό. Και τώρα κάποιο, κάποιο νομίζω, σε μια πιο παγκόσμια προοπτική. Ε, αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να διαφωνήσω για την έλλειψη ε, αρτιότητας αυτού του διτού ορισμού των τυπικών και μη τυπικών μορφών εργασίας, γιατί ε, εδώ καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος ε, ε, συμβάσεων. Και σίγουρα έχουμε μια πληθώρα νέων εργασιακών συνθήκων και εργασιακών ρυθμίσεων και πιστεύω ότι καλύπτεται με το διαχωρισμό αυτό, αυτή η πολυμορφία. Επίσης θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στις βιομηχανικές χώρες και στην Ευρώπη, κατά μέσο όρο 70% των ε, εργαζομένων έχουν ε, συμβάσει αορίστου χρόνου. Οπότε η χαρακτηριστική, η τυπική μορφή απασχόληση είναι αυτή, ε, συμβάσει αορίστου. Οπότε είναι σχετικό το βάρος των μη τυπικών μορφών εργασίας. Αλλά σίγουρα αυξάνεται όλο και περισσότερο το δικό του βάρος και το μερίδιό τους και αυτή την εξέλιξη θα πρέπει να την παρακολουθήσουμε και να την επιβλέψουμε. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι δεν είναι κατά ανάγκη όλες οι μορφές με τυπικής απασχόλησης κακές ή ε, δεν έχουν κατά ανάγκη κακή έκβαση ή δεν αποφέρουν αρνητικά αποτελέσματα. Και τέτοιου μη τυπικές μορφές απασχόλησης είχαμε ανέκαθεν. Και ένα παράδειγμα είναι ε, η προσωρινή απασχόληση. Και υπήρχαν λόγοι ε, που θεσπίστηκαν τέτοιε μορφέ απασχόληση. Η αντικατάσταση ενό εργαζόμενου, μια εργαζόμενη που βγήκε με γονική άδεια. Με άδεια μητρότητα. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δαιμονοποιούμε τέτοιε μορφέ μη τυπική απασχόληση. Έχουν κάποιο λόγο και όταν χρησιμοποιούνται ένομα είναι ευπρόσδεκτες το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές γίνεται κατάχρηση των μη τυπικών μορφών απασχόλησης ε, για λόγους ε, άσχετους με αυτούς της αρχικής τους θέσπισης. Και έχουμε ε, επιχειρήσεις που το 70% του εργατικού δυναμικού απασχολείται με μη τυπικές μορφέ επιχείρηση. Οπότε, πόσο βιώσιμη μπορεί να είναι τέτοια επιχείρηση που με τέτοιε συνθήκε οι συμβάσει απασχολεί του εργαζομένου τη. Επίση, είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλες αυτές τις πόρειες, τις διαδρομές. Δηλαδή, όταν ε, αρχίζει κανείς και απασχολείται, σε ποια φάση θα απασχοληθεί με τέτοια μη τυπική μορφή απασχόληση και πώς αυτό ε, υπονομεύει τις μεταγενέστερες πιθανότητες ε, για επαγγελματική εξέλιξη. Οπότε να δούμε μήπως μια τέτοια μη τυπική μορφή απασχόλησης είναι φαλτήριο για μια γενικότερη υποβάθμιση της. Ευχαριστώ με αυτή την τελευταία απάντηση να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες του πάνελ για τις συνεισφορές τους. Τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε κάποια συμπεράσματα. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στην Έρικα. all, uh, as deputy director, you are permanently. Ως ε, υποδιευθύντρια βεβαίως έχετε συνεχώς ε, πίεση γιατί έχετε όλες αυτές τις έχετε όλες αυτές τις δουλειές να διευθύνετε. Βεβαίω το θέμα ακριβώ ε, των ποιοτικών συνδικών εργασία είναι κάτι το οποίο απασχολεί την Κομισιόν, του κοινωνικού εταίρου, στο εθνικό επίπεδο, στο παγκόσμιο επίπεδο και βεβαίω ε, κολακευόμαστε, αλλά είναι και πρόκληση οπωσδήποτε αυτό το οποίο λέει ο Στεφάν, ότι πρέπει να γίνεται αυτή η έρευνα συχνότερα. Ναι, την κάνουμε κάθε πέντε χρόνια και λόγω του ότι εμείς είμαστε μικροί θα έλεγα ως ίδρυμα και ως Think Tank δεν μπορούμε να υποσχεθούμε κάτι. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποσχεθούμε, οι συνάδελφοί μου αλλά και η Ματέν και ο Ζώος, είναι ακριβώς οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τις συνθήκες εργασίας, είναι οι επαφές με τον ILO, τον ΩΣΑ, αλλά και με τα κράτη-μέλη με τις στατιστικές υπηρεσίες και με όσους παρέχουν έρευνες στο εθνικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα τα οποία πρέπει να δούμε και να συνδέσουμε και υπάρχει ακριβώς περιθώριο βελτίωσης και ανάπτυξης. Επίσης ήταν σαφές σήμερα ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαρες τάσεις στην Ευρώπη, υπάρχουν συγκλήσεις και αποκλήσεις ταυτόχρονα και μας ενθαρρύνατε να ψάξουμε βαθύτερα και βλέπουμε κάποια δεδομένα. 85% των εργαζομένων στην Ευρώπη είναι πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι. Το διάστημα και λέω μωρέ μπράβο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω, δηλαδή ακόμα και από τη Γερμανία 20% των εργαζομένων όμως σημαίνει ότι έχουν άσχημες δουλειές που δεν τους ικανοποιούν. Οπότε θα το εξετάσουμε αυτό σε μεγαλύτερο βάθος, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις ανισότητες που ανακαλύψαμε, για τις δουλειές χαμηλής ποιότητας, υποπίεση. Από την άλλη οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν και βελτιώσεις. Να τονίσω ένα έβριμα. Για όταν μιλάμε για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, υπάρχει μια μικρή αύξηση, αν δούμε όλους τους δείκτες μαζί, αλλά το είπε και ο Στεφάν, υπάρχει μια εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, υπάρχει πίεση, δουλειές χαμηλής ποιότητας. Ε, θα αναφέρω κάποιες ομάδες όπου θα κάνουμε πιο συγκεκριμένες αναλύσεις τα επόμενα έτη. Πρώτα απ' όλα σχετίζονται με το θέμα του φύλου, υπάρχει η διάσταση του φύλου και υπάρχει πρόβλημα ίσης ε, αντιμετώπισης στην αγορά εργασίας και όσον αφορά τις καλές θέσεις εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επίσης θα εστιάσουμε στο επίπεδο των κρατών μελών γιατί είναι πολύ ετερογενή τα αποτελέσματα και πιθανώς με κάποια δεδομένα από άλλες πηγές. Να δούμε και το περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω η Μαρίτα εδώ, η αντιπρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης, είπε πως η ετερογένεια ε, υπάρχει κυρίως στο ε, περιφερειακό επίπεδο. Μπορεί να το διαβάσατε, ο Γενικός Διευθυντής του ΑΕΛΟ ε, είπε πως ε, τα αποτελέσματα του λαϊκισμού στην Ευρώπη και στη ΣΥΠΑ οφείλονται στο ότι δεν έχουμε εμείς αποτελέσματα. Οπότε πρέπει να συνδέσουμε την κοινωνική ασφάλεια, την ευελίξ ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη και η συνδεσιμότητα αυτή που ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής, ο Μισελ, είναι στο πρόγραμμα μέσω του κοινωνικού πυλώνα και για να είμαι ειλικρινής, ε, είναι καλές οι λέξεις, αλλά πρέπει να γίνει κάτι περισσότερο. Και βεβαίως εμείς ε, χαιρόμαστε για το ότι ήδη ακριβώς υπάρχει αυτός ο πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων και συνεισφέρουμε. Θα σας κάνω μια ανάλυση που θα κάνουμε το 2017 και 2018 και θα προσκαλέσουμε ειδικά τον τομέα των πανεπιστημίων, Francis Green, Dominique, τους συναδέλφους από τον ΑΕΛΟ και τον ΟΣΑ, για να κάνουν ακριβώς την ανάλυση των δεδομένων μας, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αξίζει να επαναληφθεί είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τον ΑΕΛΟ και να δούμε τα δεδομένα με τις ε, ΗΠΑ, Νότια Κορέα και ίσως και Λατινική Αμερική κατόπιν θα μπούμε σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειες όσον αφορά τις εργαζόμενες διαφορετικής ηλικία, όπως έγινε και στο προηγούμενο πάνελ, να αναλύσουμε τις συνθήκες εργασίας και βεβαίως την εμπλοκή των εργαζομένων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους ε, για να αναπτυχθεί το επίπεδο εταιρεία και στρατηγική πολιτική. Αυτοί νομίζω είναι οι δύο πυλώνε καλύτερη πολιτική στο μέλλον. τέλο. θα κοιτάξουμε βεβαίω την υγεία των εργαζομένων, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε δύο υπηρεσίε βεβαίω για όσα που ασχολείστε περισσότερο με την ασφάλεια και την υγιεινή όπως αντιλαμβάνεστε. Και θα κάνουμε και μία ανάλυση, την ανέφερε η Μπάρμπαρα όσον αφορά το καθεστώς απασχόλησης και τι σχέση έχει και τι μπορούμε να μάθουμε και τέλος 17 αναφέρθηκε ε, ο συνάδελφος ότι έχουμε κάποιο πρόγραμμα για να δούμε ακριβώς την βιώσιμη εργασία και θα γίνει και μία μελέτη σκόπιμότητας να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι δείκτες για την ποιότητα εργασίας και βεβαίως θα καλέσουμε και τους ε, πανεπιστημιακούς ε, στον τομέα. Τέλος το 2018 θα δούμε τα διάφορα σετ δεδομένων που έχουμε. Έχουμε την έρευνα συνθήκων εργασίας και την έρευνα ποιότητας ζωής ε, που κάνουμε αυτή τη στιγμή και εστιάζει στους πολίτες. Όπως ξέρετε, εστιάζει στους εργαζόμενους η άλλη έρευνα και θέλουμε ακριβώς να έχουμε όλα αυτά τα δεδομένα για την συμφιλίωση ακριβώς ε, της εργασιακής και της προσωπικής ζωής. Και ελπίζουμε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Τέλος, θα δούμε και ως ομάδα τον ρόλο των κινήτρων για να μείνουν οι εργαζόμενοι περισσότερο χρόνο στην εργασία, αλλά και να περιλάβουμε και άλλα σετ δεδομένων, καθώς βεβαίως ε, στρατηγικά ο μεγαλύτερος χρόνος εργασίας έχει σημασία και χρειαζόμαστε και περισσότερα στοιχεία για να διασφαλίσουμε ότι αυτοί που χαράζουν την πολιτική θα εφαρμόσουν αυτά τα ευρήματα. Και είναι σημαντικά τα δεδομένα, αναφέρθηκε, το πλαίσιο μας φαίνεται ότι ακριβώς ε, είναι ιδανικό για όσους χαράζουν πολιτική. Τέλος, ανέφερα αυτό το λεγόμενο Survey Mapping Tool, το εργαλείο καταγραφής των ερευνών. Όλα μας τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. δεν ήταν διαθέσιμο σε 9 το πρωί, τώρα όμως είναι διαθέσιμο, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα, έχουν ανέβει όλα και θα χρησιμεύσουν ειδικά σε think tank, σε πανεπιστήμια, τους οποίους προσκαλούμε να τα χρησιμοποιήσουν και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλους τους φορείς. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να ζητήσω για την επόμενη φορά είναι ένας καφές. Γιατί η ισορροπία αυτή τη ζωή, με την εργασία το απόγευμα κάπως υποφέρει χωρίς καφέ. Αλλά τέλος πάντων δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητέ και ευχαριστώ και του συναδέλφους μου και την ομάδα που οργάνωσε την εκδήλωση και το γραφείο μας των Βρυξελών. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον και βεβαίως ε, καλό σας βράδυ. Ναι, ναι και τους διερμηνείς, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερμηνεία που μας χρησιμεύσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Have a nice evening. Καλό σας βράδυ. Και τα λέμε σε λίγο. Ναι. Βιστό. Ah, I forgot Matthew, our dearest cartoon. Α, ah, τον Μάθιου ξέχασα που έκανε τα σκίτσα. Τον είδατε. Έκανε πολλέ πολλές εικόνες. Ναι, ναι, θα το ανεβάσουμε στη σελίδα μας.